Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Σας καλωσορίζω όλους. Το πρώτο σημείο είναι η αποδοχή της ημερήσιας διάταξης. Δεν έχει υπάρξει κάποια πρόταση τροποποίησης από οποιονδήποτε συνάδελφο για να υπάρξουν αλλαγές Με την αφορμή αυτή θα ήθελα να πω ότι ο χρόνος που θα δώσουμε στα μεμονωμένα σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι σχετικός βέβαια, αλλά επειδή έχουμε πολλά θέματα είναι δύσκολο να είμαστε επακριβείς. Γι' αυτό παρακαλώ να ανταλάβετε υπόψη σας αυτά τα οποία λέγονται στον προγραμματισμό. Το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου, δεν υπάρχει όμως κάτι που να έχω να σας πω, οπότε περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι η συνέχεια της συζήτησης για τον Γενικό Κανονισμό 2014-2020. Ενθυμίστε ότι τους τελευταίους μήνες εμείς συγκεντρώσαμε την προσοχή μας σε διάφορα σημεία του διακανονιστικού πλαισίου για τη συγκεκριμένη περίοδο. Όλα αυτά τα θέματα, τα οποία συνδύονται με το νέο διακανονιστικό πλαίσιο, έχουμε εισηγητές από την Επιτροπή των Περιφερειών. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται η συζήτηση ενός νέου κανονισμού, θα δίδουμε 10 λεπτά στους συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειών. Και για τον γενικό κανονισμό η συγητής είναι η Κατιούσα Παρίνη αλλά δεν μπορεί να είναι παρούσα. Έχουμε όμως τη Mercedes Μπρέσο, την πρόεδρο, και θα ξεκινήσω λοιπόν δίδοντας το λόγο στη Mercedes. Όχι πάνω από 10 λεπτά παρακαλώ, ελπίζω να μπορέσετε να περιοριστείτε λίγο και μετά θα ακούσουμε πρώτα τους εισηγητές και μετά τους υπολείπους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν το λόγο. Η κυρία Μπρέσο, πρόεδρε, συνάδελφοι, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να πάρω το λόγο στην Επιτροπή σας αντιπροσωπεύω την εισηγήτρια, αλλά για μας το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δική σας απόφαση είναι πολύ σημαντική και αυτό δείχνει και η παρουσία μου εδώ ως Προέδρο. Εμείς ήμασταν το πρώτο κοινοτικό όργανο που εκφραστήκαμε γύρω από το λεγόμενο νομοθετικό πακέτο και ε, θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όσο νωρίτερα πετύχουμε κάτι τέτοιο, πόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις γνωμοδοτήσεις των νομοθετών. Ξεκινώ ε, αναφερόμενο στην ουσία της εκθέσεως, την οποία υιοθέτησε η έκθεσή μας κοτέρ, όπως λέγεται, τον προηγούμενο, στις αρχές του προηγούμενου Μαρτίου ξέρετε ότι ώσπου να φτάσει στην Ολομέλεια στις αρχές Μαΐου δεν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Το πρώτο θέμα είναι η αρχή της εταιρική συνεργασίας και η λεγόμενη πολυεπίπεδη governance, η διακυβέρνηση. Ξέρετε ότι αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας και ζητάμε την πλήρη εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επεξεργασία, στην διαπραγμάτευση, στην εφαρμογή και στην αναθεώρηση των αποφάσεων, των συμβάσεων, των κοινών στρατηγικών κτλ. Θεωρούμε άδικη, αν θέλετε, την ταύτιση των τοπικών και περιφερειακών ερχών με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με την κοινωνία των πολιτών δεν είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό οι περιφέρειες της Ευρώπης προτείνουν την πλήρη συνεργασία τους στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης εταιρικών σχέσεων. Ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις, πολλές θα έλεγα στην Ευρώπη, όπου οι περιφέρειες στο εσωτερικό του κράτους είναι συνδιαχειριστές και μάλιστα μερικές φορές και ε, ε, χρηματοδότες των προγραμμάτων. Η Επιτροπή λοιπόν των Περιφερειών επιμένει στην πολυεπίπεδη αυτή governance. Ε, θα εκφράσουμε την άποψή μας σε έφθετο χρόνο και με τον κώδικα συμπεριφοράς για την εταιρική σχέση και θα αναλύσουμε σε βάθος το σύνολο των προγραμμάτων που έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ελέγξουμε ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εμπλέκονται παρκώς. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ είναι η συγκέντρωση και η ολοκλήρωση των ταμείων στο λεγόμενο κοινό στρατηγικό πλαίσιο ταμείων. Υπάρχει ανάγκη να συγκεντρωθούν, να στοχοποιηθούν τα διαφορετικά ταμεία σε ένα περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων σε σχέση με την Ευρώπη του 2020. Ζητάμε όμως, όπως και στα πλαίσια του εγγράφου που σας καταφέσαμε, μια μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των προτεραιοτήτων αυτό και γι' αυτό προτείνουμε την κατάργηση των ελαχίστων ορίων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ανάμεσα στις θεματολογίες της Ευρώπης του 2020. Οι περιφέρειες θα πρέπει να επιλέγουν τις προτεραιότητες. Τέλος, πιστεύουμε ότι για να είναι αποτελεσματική η πολιτική αυτή θα πρέπει να σέβεται τους περιφερειακούς εταίρους. Οι θεματολογίες δεν μπορούν να καθορίζονται μόνο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τώρα, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε ακόμα σε ένα επίπεδο, ε, θα έλεγα, ε, κειμένου εργασίας. Εκφέρουμε μία γνωμοδότηση ζητώντας να υπάρξει ουσιαστικό συντονισμός ανάμεσα στο ταμεία, ανάμεσα στο ΦΕΔ, ανάμεσα στα ταμεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο κτλ. Και ζητάμε να υπάρξει μια πραγματική δυνατότητα εφαρμογής και πραγμάτωσης των συγκεκριμένων αυτών προγραμμάτων. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να είναι παράρτημα του κανονισμού και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο έκρησης μέσω της συναπόφασης και από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτο θέμα είναι η πολιτική θα έλεγα την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε σχέση με την αρχιτεκτονική της λεγόμενης συνοχής. Εμείς ε, έχουμε αναφερθεί στην κατηγορία των ε, εν μεταβάση περιφερειών που καλύπτουν ακριβώς λόγω των πολλών αλλαγών όλο και περισσότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάποιες αναπτυγμένες περιοχές άνω του 90% πέφτουν ε, λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις ε, παραγωγικές περιοχές οι οποίες υφίστανται τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η κρίση οικονομική εν πολλής δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση του κατακεφαλήν ΑΕΠ των θα έλεγα κινητήριων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω των δυσκολίων τις οποίες δημιουργεί η κρίση σε αυτούς που είναι ευάλωτοι στον διεθνή ανταγωνισμό. Εμείς λοιπόν μας απασχολεί η κατηγορία αυτή των υπομετάβαση περιφερειών και παρακολουθούμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο με ενδιαφέρον. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στις δύο επιτροπές και η Περιφερειακή Επιτροπή του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Προϋπολογισμών ακολουθούν μερικές φορές διαφορετικές κατευθύνσεις γύρω από το θέμα αυτό. Τέταρτο θέμα η αιρεσιμότητα και οι επιδόσεις. Δεν υπάρχει ομοφωνία σε σχέση με την αιρεσιμότητα στην Επιτροπή Περιφερειών. Εμείς έχουμε αρνηθεί την λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θεωρούμε ότι οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές και η ίδια η πολιτική συνοχή είναι όμοιροι πλέον και τιμωρούνται από αυτήν την σταθεροποιητική μόνον πολιτική και την έλλειψη αντισταθμισμάτων από πλευράς των κρατών μελών που απλά θέλουν να μειώσουν το, το έλλειμμα. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια επιτάχυνση της εκ των προτέρων ε, προσπάθειας ορισμού της αιρεσιμότητας. Κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σας ζητώ επίσης να εξετάσετε τις τροπολογίες για το παράρτημα 4, ιδιαίτερα την δική μας τροπολογία υπαρίθμη 63 η οποία προβλέπει 20 παρεμβάσεις απλούστευσης σε σχέση με τους προτινόμενες ρυθμίσεις. Έχουμε επεξεργαστεί πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι ότι η σύγκληση και η συνοχή έχουν προτεραιότητα και όχι η απόκληση και η διαφοροποίηση και δεν θα πρέπει να τιμωρούμε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα. Θεωρούμε ότι η ευαισθημότητα δεν θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί με ένα σύστημα οικονομικών κυρώσεων, ούτε και με ένα σύστημα αμοιβών αν θέλετε, σε σχέση με τις λεγόμενες επιδόσεις performance. Πρώτον, η αμοιβή των καλυτέρων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποια προβλήματα και δεύτερον οι στόχοι οι οποίοι πολλές φορές είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Είμαστε όμως υπέρ ενός αποθεματικού ευελιξίας. Ένα πέμπτο σημείο, απλούστευση των διαχειριστικών κανόνων και των ελεγκτικών κανόνων. Εμείς θεωρούμε ότι ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική απλοποίηση των προβλέψεων. Η αίσθηση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πρόταση στην ουσία προβλέπει απλοποιήσεις μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυξάνει την περιπλοκότητα του ελέγχου για τις εθνικές αρχές και τις τοπικές αρχές. Έχουμε επίσης αμφιβολίες και για την Υπουργική Αρχή Πιστοποίησης η οποία τίνει να επιβαρύνει ένα σύστημα ιδιαιτέρως περίπλοκο και σε επίπεδο εκ ελέγχων και σε επίπεδο διαχείρισης περιφερειακής. Υπάρχει μία πρόταση απλούστευσης από δικής μας πλευράς την οποία θα ήθελα να σας καλέσω να εξετάσετε προσεκτικά γιατί πολλές από τις περιφέρειές μας είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τα ποσά αυτά και γι' αυτό έχετε τη δυνατότητα να τα ελέγξετε σωστά. Τώρα, η εδαφική ενότητα, θα έλεγα, της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Ένα θέμα που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι η εδαφική διάσταση. Από αυτή την άποψη χαιρετίζουμε ε, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ των τοπικών δράσεων και των ολοκληρωμένων επενδύσεων. Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την περιπλοκότητα των τρόπων επίτευξης των δύο προηγούμενων στόχων. Είμαστε επίσης υπέρ του νέου Urban, έχοντας όμως την ανησυχία ότι υπάρχει ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός στόχων από τη μία όλες οι πολιτικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στις, ατικές, στις αστικές περιοχές ε, κατά κάποιο τρόπο σπάνε την τακτική που έχουμε σε σχέση με τη συγκέντρωση των στόχων. Ζητάμε λοιπόν εδώ την προσοχή σας. Θέλουμε επίσης ε, να χρηματοδοτούνται και στα πλαίσια ε, των αναπτυγμένων περιοχών οι υποδομές οι οποίες χρήζουν ανακαινήσεων. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε επίσης τη συνέχιση των πολυπεριφερικών προγραμμάτων που βασίζονται σε κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει εδώ να τεθεί το θέμα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής όπως την ονομάζουμε στα πλαίσια της συνοχής και ελπίζουμε να υπάρξει και ειδική αντιμετώπιση για τις υπερπεριφερικές ζώνες. Συμπερασματικά, λέει η κυρία Μπρέσο, σας ζητώ να διαβάσετε τη γνωμοδότησή μας. Προτείνουμε 60 περίπου τροπολογίες στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για σας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε όπως είπαμε υπέρ και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεν έχουμε τον κύριο Σίμιτσεκ μαζί μας, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο αν θέλετε είναι εκτός του θέματος που συζητάμε τώρα, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Είμαστε υπέρ της ένταξης στην πολιτική της λεγόμενης συνοχής ε, του κοινωνικού ταμείου φυσικά, στα πλαίσια του κοινού στρατηγικού πλαισίου και είμαστε και υπέρ της περιφερικοποίησης ε, του ταμείου αυτού λόγω του ρόλου των περιφερειών ε, σε κάποιες χώρες είναι ήδη περιφερικοποιημένο το ταμείο αυτό και πρέπει να προχωρήσει και εκεί που δεν είναι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, uh, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω τώρα το εξή να ακούσουμε πρώτα τις αντιδράσεις των μελών στα ε, ε, όσα μας είπατε. Πρώτα από τους δύο εισηγητές, η κυρία Κρέλ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα και να μπω στα θέματα που είχαμε για σήμερα προβλέψει στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ καταρχάς ε, ιδιαιτέρως και ειλικρινά την κυρία Μπρέσο και για το γεγονός ότι ήρθε αυτοπροσώπος στην Επιτροπή μας. Πολύ μεγάλη μας τιμή με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, νομίζω, έχουμε και εμείς αντίστοιχα προβλήματα εντοπίσει. Τα ίδια θίγουν και εκείνοι. Ας πούμε η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ή ε, τι γίνεται με τις συμβάσεις εταιρικέ. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Επίσης το θέμα της απλούστευσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λίγα είναι τα πράγματα που μπορεί να διαφέρουμε σε αποχρώσεις όμως στις απόψεις μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο που έχουμε εδώ την Επιτροπή Περιφερειών και στο μέλλον να κάνουν και ισχυρό λόμπι παρακαλώ στα κράτη-μέλη να πιέζουν γιατί εκεί είναι το επόμενο στάδιο και η επόμενη βαθμίδα για να προετοιμάσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο οι περιφέρειες εκεί καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο πλέον κρατών μελών. Σήμερα είχαμε συμφωνήσει να συζητήσουμε ορισμένα θέματα που αναφέρετε και εσείς που είναι η ανάπτυξη, η αστική, η απλούστευση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ε, διασταυρούμενη χρηματοδότηση, το περίφημο multifund, ε, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Είχαμε αναβάλει την αστική ανάπτυξη, γιατί θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα παρευρέσει και το Γιάνν Όλμπρεχτ. Και φαίνεται και από το έγγραφο εργασίας ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένη η υπόθεση αυτή και με το γενικό κανονισμό και με τον άλλο κανονισμό για το ειδικό ταμείο. Γι' αυτό έπρεπε να είναι παρόντες και οι τρεις συζητητές και να είναι σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία. Στόχος όλων είναι να αυξήσουμε την ανάπτυξη των πόλεων, ιδιαίτερα ως προς την αηφορία και τη βιωσιμότητά της. Γι' αυτό κονίσαμε και μια κοινή πρόταση να δίνουμε τη δυνατότητα στις πόλεις να αναπτύσσουν δικά τους έργα, προγράμματα, ενδεχομένω και με συνολική χρηματοδότηση, αλλά αυτό είναι θέμα του Γιάνν Όρμπρεχτ και θα το προτείνει για το ταμείο του. Πάντως έχουμε συμφωνήσει ότι το 5% που είναι η ελάχιστη χρηματοδότηση ως συντελεστής για την αστική ε, η ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου να είναι δεδομένη. Σε περίπτωση που πραγματικά έχουμε τέτοια προγράμματα και σχέδια από τις πόλεις. Να έχουν τη δυνατότητα στις περιφέρειες οι πόλεις να αναπτύσσονται και με τις αντίστοιχες στρατηγικές και μέσα που προβλέπουν οι εκάστοτε κανονισμοί. Το ITIS για παράδειγμα, αλλά Κάπου το έχουμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα και είπαμε ότι είναι δύσκολο αυτό που προτείνεται ως βελτίωση. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε ως ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ο κατάλογος των 300 πόλεων που θα πρέπει να συνοδεύεται και να φωτίζεται και από μια εταιρική σύμβαση εδώ. Διατηρούμε πολύ μεγάλες επιφυλάξεις έχει άραγε καμιά ευρωπαϊκή υπεραξία αυτό ή προστιθέμενη αξία για τις ίδιες πόλεις. Υπάρχει το URB Act, το EuroCities, υπάρχουν προγράμματα που συνεργάζονται πόλεις για ανταλλαγές ε, εμπειριών, πληροφοριών, βελτιστών πρακτικών ε, για ευρωπαϊκά θέματα. Δεν χρειάζεται νομίζω και άλλος ένας κατάλογος. Είναι άχρηστη επιβάρυνση κατά τη γνώμη μου και για τις συμβάσεις αυτές ε, από την αρχή εκ των προτέρων χωρί κάποιος να ξέρει ποια έργα είναι αυτά και ποια σχέδια να αποφασιστεί ένας οριστικός κατάλογος 300 πόλεων όχι. Θα θέλαμε λοιπόν να παραμείνουν οι παλιές δομές, τα υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας των πόλεων και το 5% των διαρθρωτικών πόρων να αφιερωθεί σε πραγματικά νέα έργα στις πόλεις. για τις αστικές και περιαστικές περιοχές βεβαίως και καινοτόμα ε, μέτρα που θα πρέπει να προωθηθούν. Έτσι τονίζεται και η λεγόμενη εδαφική διάσταση της αστικής ανάπτυξης και ακριβώς αυτό είναι το θέμα που έχουμε λάβει την εντολή ως κοινοβούλιο να το προωθήσουμε και ε, με τις νέες ρυθμίσεις για την εδαφική συνοχή στις συνθήκες. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι βεβαίω θα χρειαστεί και περαιτέρω συζήτηση σε λεπτομέρειες. Επί τη ουσίας θα τα ξανασυζητήσουμε και αυτό είναι περισσότερο ε, δουλειά του Γιάνν Όλμπρεχτ που είναι εισηγητή για αυτό το ταμείο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να έχουμε ένα άξονα προτεραιότητας για αστική ανάπτυξη και να συντονίσουμε διάφορες θεματικές ενότητες και άξονες προτεραιοτήτων και πολιτικής. Θα τα ξαναδούμε αυτά με τους συγητές και ιδιαίτερα με τον Γιάνν Όλμπρεχτ. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της απλούστευσης στη διαχείριση των πόρων από τα διαφορετικά ταμεία. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια. Βεβαίω είναι σωστό ότι η συνένωση των πέντε ταμείων σε ένα γενικό κανονισμό με την ίδια μέθοδο για την αξιολόγηση, την εκτίμηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο βοηθάει φυσικά. Στην αρχή θα υπάρξουν κάποια προβλήματα προσαρμογής, αλλά μακροπρόθεσμα ε, θα βοηθήσει. Έχει δίκιο η κυρία Μπρέσο, στην αρχή ενδεχομένως μπορεί να έχει λιγότερα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ε, δυσκολευτούν. Στη συνέχεια όμως θα είναι χρήσιμο μέσο γιατί αν προετοιμαστεί σωστά και εφαρμοστεί σωστά θα είναι πραγματικά απλούστευση για όλους τους ε, δικαιούχους. Θα πρέπει να ρωτήσουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει προετοιμάσει σωστά την ηλεκτρονική συνοχή, το e-cohesion, εάν υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση ανάγκης να επανέλθουμε και στο χαρτί, εν περιπτώσει, όχι όλα ηλεκτρονικά, γιατί δεν έχει και το τελευταίο σωματείο δυνατότητα ηλεκτρονικής ε, διεκπαιρέωσης και επεξεργασίας. Πάντως, καλό είναι να προτείνουμε στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν, γιατί η μακροπρόθεσμα θα είναι ακριβώς ο καλύτερος τρόπος και ο πλούστερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι θετική η συμβολή αυτή προς την κατεύθυνση της απλούστευσης. Επίσης, είναι γεγονός ότι πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια που υπάρχει. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε αν υπάρχουν συστήματα που ανταποκρίνονται και στην προστασία των δεδομένων. Δηλαδή ηλεκτρονικές υπογραφές που να αναγνωρίζονται και τέτοια στοιχεία ασφαλείας που να προστατεύονται κάποιες πληροφορίες ότι δεν θα συμβεί τίποτα στραβό. Αλλά αυτά θα τα δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα θα μας τα εξηγήσει στο επόμενο διάστημα τις επόμενες εβδομάδες. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να μπει στο γενικό κανονισμό και τελευταία τεχνική λεπτομέρεια. Κάποιο ρώτησε και γιατί γίνεται με τι δυνατότητε πολλαπλής χρηματοδότησης, το MultiFunds, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρόντισε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στο, στο νέο κανονισμό, ενώ στο σημερινό αυτό δεν γίνεται και πρέπει να γίνει διάκριση κάθε φορά ανάμεσα στα διάφορα έργα, τα hard και soft, ε, ως προς τις επενδύσεις. Τώρα προσπάθησαν να αλλάξουν προσέγγιση. Δυστυχώς όμως αυτή η προσέγγιση δεν φτάνει μέχρι το επίπεδο του έργου αυτού καθ' αυτού, μόνο μέχρι τους άξονες προτεραιότητας. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να κάνει πρόταση. Για να φτάσουμε μέχρι το επίπεδο του έργου κάθε φορά, όχι. Ε, γιατί ε, αυτό είναι το καλύτερο και έχει το περισσότερο νόημα για τους ενδιαφερομένους. Αλλιώς θα πρέπει ο κάθε διαχειριστής του έργου να το διαχωρίζει ε, στα ταμεία. Δεν ξέρω μήπως είναι αυτό επιπλέον δουλειά και επιβάρηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω και πρόκληση, αλλά αξίζει τον κόπο να ανταποκριθεί σε αυτή για να φτάσουν τα θετικά αυτή της προσέγγισης ε, και στους τελικούς δικαιούχους. Εκεί και το θέμα της διασταυρώμενης χρηματοδότησης αυτό στο multifund. Εάν πραγματικά υπάρξει τέτοια ρύθμιση μέχρι το επίπεδο του project, δεν χρειάζεται τελικά μάλλον η διασταυρούμενη χρηματοδότηση, γιατί επικαλύπτεται ε, με το προηγούμενο ή το ένα καταργεί το άλλο. Σε περίπτωση όμως που δεν καταφέρουμε το ε, multi να το φτάσουμε μέχρι το έργο, ε, Ας το περιορίσουμε στο 10% όπως προτείνεται αυτό. Αυτά τα ολίγα ως ε, εισαγωγή και σταματώ εδώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε αργότερα τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριος Βανίστερόι. Ε, αν δεν θέλεις, να ακούσουμε τους άλλους. Φιλελεύθεροι. Ποιος θέλει από τους φιλελευθέρους ως συγητής Κιώδης. Uh, Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να επιλύσουμε είναι η κατάρτιση των συμφωνιών συνεργασίας. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή ποια είναι η πραγματική συμμετοχή της περιφέρειας, διότι διαφέρει πάρα πολύ. Πρώτη φορά καταρτίζεται ένα τέτοιο έγγραφο και το βασικό θέμα για το Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι ότι εάν καταρτιστεί μέσα σε μία χώρα ε, που είναι η συνήθις αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους μέλους, τότε το κράτος μέλος φροντίζει ε, σύμφωνα με τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες να εμπλέξει και την περιφέρεια και να καταρτήσει τα αναγκαία έγγραφα. Επίσης, ή διαφορετικά επιμένουν εκ του παραλίλου η περιφέρεια πέραν των εκλεγμένων εθνικών ε, εκπροσώπων, ε, των βουλευτών δηλαδή, ε, να καταρτήσουν έγγραφα, ένα πλαίσιο και μία συμφωνία συνεργασίας. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν προτού υιοθετήσουμε τον κανονισμό αυτό. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει εδώ άλλος ε, εισηγητής. Θέλετε να μιλήσετε εν ονόματι των Πρασίνων, ο Φρονσουά Αλφόνς. Με συγχωρείτε. Ε, Δύο-τρεις σκέψεις. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειών για αυτή την εργασία, την οποία θεωρώ εξαιρετική. Συμφωνούμε με τις ανησυχίες, διότι καταρχήν Όντως ε, αισθανόμαστε στο διάβημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη θέληση να βελτιωθεί η κατάσταση, να γίνει μια καλύτερη πολιτική περιφερειακή, αλλά ε, είναι μια πολύ κατευθυνόμενη διαδικασία και δεν βλέπουμε μία κατάρτιση ενός επταετούς προγράμματος ανάπτυξης με ε, ανταλλαγές και συζητήσεις με τους εταίρους και διαπιστώνουμε ότι στις ε, πρακτικές διατάξεις ε, δεν υπάρχει τονισμός της πτυχής της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να ενισχύσουμε ενισχυθεί. Επίσης όσον αφορά την επίδοση εμείς θεωρούσαμε πάντοτε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία και όχι βαθμολόγηση ε, των ανθρώπων με τον οποίο λειτουργούν και ε, πιστεύω ότι εδώ αντιμετωπίζονται σωστά η περιφέρεια, πολλά πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, πολλά μπορούν να γίνουν, ε, κάτι που είναι σήμερα προτεραιότητα αύριο μπορεί να μην είναι, προκύπτουν νέα θέματα Χρειάζεται δηλαδή μία ευελιξία έναντι των επιδόσεων οι οποίες βαθμολογούνται και είναι αφιλεγόμενες. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο στηρίζουμε και ιδίως όταν μιλάμε για τον ο χώρο ε, της ε, αποτελεσματικότητας δέχεται ε, να αφήσουμε ορισμένες προτεραιότητες κατά μέρος, να επιλέξουμε άλλες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τις θεματικές προτεραιότητες όπως ελέγχθη ή να τις συγκεντρώσουμε σε κεφάλαια για να εξετάσουμε πιο ευρία θέματα και κεφάλαια που θα μπορέσουν να οργανωθούν και να διεκπαιρεωθούν πιο εύκολα. Το τρίτο που τονίζουμε είναι η απλοποίηση. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο διότι χρειάζεται αυτή η συνειδητοποίηση η οποία μπορεί να προέλθει από τις θετικές διατάξεις αλλά δεν είναι μονόδρομος. Δεν πρέπει απλώς να απλοποιήσουμε τη ζωή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και των επιτόπου και επειδή ε, εγώ είμαι νησιώτης στα νησιά υπάρχουν μικροί φάκελοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιες γραφειοκρατίες σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να απλοποιήσουμε ε, και να προτείνουμε λύσεις εις τους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο στα ελεγκτικά όργανα. Ευχαριστώ. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επισημάνω και πάλι ότι αυτό το οποίο συζητάμε εδώ είναι αφενός την παρουσίαση ε, ε, ε, του Γενικού Κανονισμού από την Επιτροπή Περιφερειών μαζί με την εισηγήτρια και ε, συγχρόνως τη συζήτηση της ε, ε, αστικής διάστασης και την μη δυνατότητα μεταφοράς των πόρων και παρακαλώ την Κονέλια Ένστ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να παρέμβω εδώ εν ονόματι της Ηνωμένη Αριστεράς ε, και ευχαριστώ την Επιτροπή Περιφερειών διότι πιστεύω ότι αυτό κάπως μας καθησυχάζει το να βλέπουμε τόση συνένεση και αποδοχή των θέσεών μας και βλέπουμε ότι αξίζει να τα προωθήσουμε. Αναφέρομαι εδώ εις ε, τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατική φράση και πρέπει να τη στηρίξουμε. Ε, γι' αυτό πρεσβεύουμε σαν Ηνωμένη Αριστερά. Θα μπορούσαν όμως οι περιοχές αυτές να είναι θύματα του ότι οι θέσεις τους δεν αρέσουν σε κανένα και πρέπει να οξύνουμε ή να ενισχύσουμε τουλάχιστον ε, την ε, πτυχή αυτή. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς επί του δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερον, από πλευράς των, ε, της Επιτροπής ε, Περιφερειών βλέπω ότι η αιρεσιμό της ε, μας βρίσκει σύμφωνους, χρειάζεται μία πολιτική όπου τα κράτη δεν θα τιμωρούνται ή θα χρειαστεί να πληρώσουν για συγκεκριμένες περιοχές και δεν θα μπορεί κανείς να παρακάμψει και τις διατάξεις διότι τότε μπορεί να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και εδώ αναφέρομαι ε, στα συγκεκριμένα παραδείγματα ε, σχετικά με την συνοχή. Ε, αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά είναι να δούμε τι από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σχετικά με την κυρία Κρέλ και την ανάπτυξη των πόλεων. Πρέπει να δούμε ποια προγράμματα θα στηρίξουμε, δηλαδή τι θα γίνει με την ε, πολεοδομική ανάπτυξη, αν θα υπάρχει δικτύωση, αν θα υπάρχει προώθηση, ε, θα πρέπει να υπάρξουν νέα προγράμματα Ποια όμως, δεν ξέρω αν είναι λογικό να βάλουμε ένα ποσοστό, να μιλάμε για 4, 5 ή 6% νέων προγραμμάτων και ίσως θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε την πρόταση της Επιτροφής Περιφερειών, να δούμε αν πρέπει να ξανασκεφτούμε την πόλη, αν πρέπει να δημιουργηθεί κάτι τελείως καινούριο, να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή την Επιτροπή Περιφερειών για να υπάρξει μια νέα διατύπωση. Ε, το 5% που αναφέρεται εδώ δεν με πείθει, όπως άλλωστε και τα επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά τη δικτύωση, υπάρχουν πολλές προτάσεις, 15-20%, ό,τι ε, αυξάνει είναι καλό, υπάρχουν λιγότεροι πόλοι και έτσι ε, καλό είναι να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις διάφορες δράσεις και αυτό ολοκληρώνει τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Ντέρεκ Βον. Για την Επιτροπή των Περιφερειών θα ήθελα να πω ότι θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι με αυτά τα οποία μας είπε η Επιτροπή Περιφερειών, οι περισσότεροι από μας. Θα ήθελα να έλθω λίγο στο θέμα της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο όλοι πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό, αλλά δεν είμαι βέβαιος για το πώς σκοπεύει να το πετύχει στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό θέτουμε κάποιες ερωτήσεις και προς την Επιτροπή Περιφερειών και την Κομισιόν. Πώς θα υπάρξει συνεργασία και επαφή ανάμεσα στα διάφορα ταμεία πώς θα ελεγχθούν τα χρήματα τα οποία θα πανώνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις καινοτομίες και για τις λεγόμενες δραστηριότητες χαμηλών εκπομπών. Και υπάρχει επίσης και το θέμα των εταιρικών συμβάσεων, συμβάσεων εταιρικών σχέσεων μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι αυτές οι εταιρικές συμβάσεις θα υπογράφονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ενώ εμείς πιστεύαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κεφάλαιο για την παρουσία στις συμβάσεις αυτές επισήμως των περιφερειακών αρχών. Λοιπόν, πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το επιδιώξει αυτό. Αυτά ήθελα να θέσω κυρίως προς την Επιτροπή των Περιφερειών. Ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το θέμα της απλοποίησης. Ξέρετε ότι ασχολήθηκε και η ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών με αυτό το θέμα. είναι η προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας ανάμεσα στη σωστή χρήση των διαθεσίμων πιστώσεων και από την άλλη να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή όχι μόνο των υπηρεσιών των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και αυτών οι οποίοι ωφελούνται από τα χρήματα αυτά. Η ισορροπία ανάμεσα στους δύο αυτούς στόχους δεν είναι προφανής. Σχετικά τώρα με την πιστοποίηση της ε, οικονομικής διαχείρισης ε, και των οικονομικών ελέγχων κτλ. Όλα αυτά είναι προτάσεις οι οποίες θα πρέπει θεωρητικά να στηριχθούν, αλλά πρέπει να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την Επιτροπή. Σχετικά με τις αστικές περιοχές τώρα και το πρόγραμμα Urban, Neurban κτλ. Ιδιαίτερα ο στόχος των 300 πόλεων που μπορεί πιθανώς να ενταχθούν στην πλατφόρμα Urban ποιος θα αποφασίσει ποιες είναι αυτές οι πόλεις και ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα ποσοστά, ποιοι είναι οι όρια αναφοράς εν πάση περιπτώσει. Επανέρχομαι στην αρχή της συζήτησής μας λοιπόν. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εμπλακούν οι ίδιες οι περιφέρειες, θα πρέπει να ορίσουν οι περιφέρειες ποιες θα είναι αυτές οι πόλεις και τι ακριβώς θα γίνει για αυτές το μέλλον. Ευχαριστώ Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συζητητέ ε, που έφεραν ε, το θέμα του Urban στη σημερινή συζήτηση. Είναι και θέμα του Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα να σας εξηγήσω τη θέση μου ως πριν μπω στις λεπτομέρειες του ΦΕΝΤΕΡ. Αυτό που έχει σημασία στο γενικό κανονισμό είναι το εξή. Υπάρχει εδώ μια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη του τις διάφορες νομικές δομές στα διάφορα κρατημέρια. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν χώρες που είναι μοσπονδία κούτι, που άλλες με ιδιαίτερη αποκέντρωση και το κείμενο θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις σε κάποια κράτη. Παράδειγμα, ο κώδικας δεοντολογίας συμπεριφοράς για τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Και είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο των πόλεων. Ε, το είδαμε και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών. Θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι η εταιρική σχέση και η σύμβαση. Πρώτα να εξηγήσουμε ποιοι είναι οι εταίροι αυτοί είναι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μήπως μιλούμε ε, για εταίρους σε εθνικό επίπεδο πλέον. Και από εκεί και πέρα στο εθνικό επίπεδο ποιοι είναι οι εταίροι αυτοί και ε, πώς συνδέεται με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της ΜΚΟ και άλλους ε, κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή πώς θα καταρτίζεται αυτή η σύμβαση και τι περιεχόμενο θα έχει, εκτός του ποιος θα την υπογράφει. Είναι πολύ επίγον αυτό. Στον κανονισμό λοιπόν για τη σύμβαση έχουμε το περίφημο κατάλογο αστικών περιοχών. Δεν θέλω να μπω στο ιστορικό από που ε, προέκυψε αυτό, αλλά ως εισηγητής προτείνω και ελπίζω να το υποστηρίξετε στην Επιτροπή το εξή. Να πούμε πρώτα ξεκάθαρα ότι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχουν μια σειρά διαφορετικών δράσεων, πολύ διαφορετικών, που θα πρέπει να υλοποιούνται στις πόλεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί όρια, ε, ποσοστά. Αλλού είναι τα όρια στα θέματα και στη θεματική συγκέντρωση, αλλά σε ό,τι φορά τους συντελεστές, τα project ε, στις πόλεις, δεν υπάρχει περιορισμός. Εξαρτάται από τη διαχειριστική αρχή. Τι εννοώ εδώ. Ε, την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τις υποδομές, τις αστικές συγκοινωνίες, ε, αναζωγόνηση των πόλεων, κοινωνική, ε, ανάπλαση, οικονομική. Δεν υπάρχουν όρια εκεί. Αλλά ως εισηγητής θα ήθελα να υποστηρίξω και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα ειδικό λεγόμενο πρόγραμμα και να εξασφαλιστεί εκεί 5% της εθνικής χρηματοδότησης του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 5% το οποίο όμως θα δίδεται πρώτα για τις λεγόμενες λειτουργούσες αστικές περιοχές. Δηλαδή, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη εδαφική διάσταση από ό,τι σήμερα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν ε, τι θέλουν να υποστηρίξουν, σε ποιες λειτουργούσες περιοχές. Δηλαδή, είναι αυτό αστικές και περιαστικές περιοχές. Ένα 5% λοιπόν θα πρέπει να αφιερώνεται εκεί και να ε, πηγαίνει αποκλειστικά σε αυτές. Με ειδική μεθοδολογία αυτό είναι και στο ITI, στη μεθοδολογία του και επίσης αυτές οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν, οι περιοχές μάλλον, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και τη γενική χρηματοδότηση που είναι στο γενικό κανονισμό. Τι προτείνω λοιπόν, ή θα προτείνω στις τροπολογίες μου. Να εγκαταλείψουμε τελείως τον κατάλογο και να πούμε απλώς τα κριτήρια σε επίπεδο σύμβαση εταιρική σχέση. Και από εκεί και πέρα κάθε κράτος μέλος θα αναλύσει τι σημαίνει 5% του ΕΤΠΑ, τι πόλεις θέλουν να υποστηρίξουν και με ποιον τρόπο μετά θα χρησιμοποιούν το ITI και ε, τη δυνατότητα της γενικής χρηματοδότησης, αλλά σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, αυτό χρειάζεται και ένα ενδιάμεσο φορέα που μπορεί να δημιουργείται σε επίπεδο ε, λειτουργούς πόλης. Υπάρχει δυνατότητα γενικής χρηματοδότησης, αλλά όχι υποχρέωση. Γιατί ορισμένες από αυτές τις περιοχές της πόλης μπορεί να μην είναι έτοιμες να επομιστούν την ευθύνη για τη συνολική χρηματοδότηση, εξού και το περίφημο 5%. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λογική συνέπεια ποια ήταν. Να μπουν στην πλατφόρμα οι πόλεις του καταλόγου, να φύγουν από τον κατάλογο. Αλλά εγώ θα έλεγα να φύγουν και από την πλατφόρμα. Γιατί αν υπάρχουν κριτήρια, θα αποφασίζει ε, ποιες είναι οι αστικές αυτές περιοχές στο κράτος και ο κατάλογος θα είναι το τελικό προϊόν, δεν θα είναι αφετηρία. Και βέβαια υπάρχει δυνατότητα ελέγχου πάντα και αξιολόγησης, αλλά αυτό υπάρχει σήμερα και λέγεται airbagged. Και στην Επιτροπή Περιφερειών. Και υπάρχει και ένωση ε, και συνεργασία πόλεων έτσι και αλλιώς. Δεν χρειάζεται νέα αστική πλατφόρμα. Υπάρχουν τα δίκτυα αυτά. Και η ιδέα που λέει 300 μεγάλες πόλεις μπορεί να ήταν η αρχική μας ε, παραδοχή, η αρχική ιδέα. Αλλά τώρα ε, συζητούμε για λειτουργούσες αστικές περιοχές που εξαρτώνται και από το μέγεθος του κράτους μέλους και από το ίδιο των δράσεων που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα δοθούν για να προαγάγουν και να ε, εθαρρύνουν τις αστικές περιοχές να συνεργάζονται και να δημιουργούν δίκτυα και να κάνουν κάτι παραπάνω για να βγαίνει τη θέμενη αξία. Αυτή θα είναι η πρόταση λοιπόν ε, η δική μου. Αλλά αν μπορώ να προσθέσω τίποτα για τη σημερινή συζήτηση ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία εδώ είναι η διασταυρώμενη χρηματοδότηση. Αλλά ε, το σύστημα ε, πολλαπλής χρηματοδότησης, αν παραμένει μόνο σε στάδιο προγραμματισμού, αυτό είναι πάρα πολύ ε, ασθενές. Αν είναι σε επίπεδο προγράμματος πάλι, παραμένει επίσης ασθενές. Θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο έργου, project. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέγει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Θα είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά αν μπορούμε το σύστημα πολλαπλή χρηματοδότησης να είναι σε επίπεδο ε, project, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πλέον έκτημα. Και η διασταυρούμενη χρηματοδότηση να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη γιατί αν θεωρούμε ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο, δεν θα πρέπει να περιοριστεί αυτό στο 5-10%, πολύ περισσότερο, να 25-30% η διασταυρούμενη χρηματοδότηση. Γιατί ε, εμείς θέλουμε να, να κάνουμε τη ζωή του κόσμου πιο εύκολη και όχι να δυσκολεύουμε τα πράγματα με τεχνητές αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην πρόταση της Επιτροπής Περιφέρειων υπάρχει κάτι πολύ επίμαχο το οποίο ανέφερε η Πρόεδρος και αυτό είναι το στοιχείο της μακροπεριφέρειας. Όταν μιλούμε για το ίδιο κράτος μέλος και συνεργασία περιφερειών, καλώς. Είναι εύκολο. Αλλά όταν είναι διασυνοριακή η λεγόμενη μακροπεριφέρεια, για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα σχόλιο μόνο. Ε, όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το λέει και η Επιτροπή Περιφερειών και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως πρόταση, είναι πάρα πολύ αυστηρή αυτή τη φορά η δέσμευση των κονδυλίων εκεί σε επίπεδο και του Κοινωνικού Ταμείου και του Περιφερειακού Ταμείου. 25%, 40% ε, μετά έχουμε ε, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την οριοθέτηση ε, στην αρχή προσημειώνουμε ε, στο ταμείο και μέχρι 80% υπάρχει δυνατότητα. Για τρεις θεματικές ενότητες ή στόχους, αλλά πρέπει να γίνει μια επιλογή. Αλλιώς στο γενικό κανονισμό θα πρέπει να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, μια ταξινόμηση ε, των θεματικών στόχων, γιατί τρεις είναι σημαντικότεροι. Δεν μπορούμε να πούμε έχουμε 11, τρεις πρέπει να διαλέξουμε. Ε, δεν είναι λογικό αυτό. Και ε, επίσης περιμένω τη συζήτηση για το κοινωνικό ταμείο, γιατί εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση. Γιατί εκεί έχουμε τη συγκέντρωση σε επίπεδο προγράμματος. Εδώ λοιπόν λέμε ότι όλα θα είναι πιο ευέλικτα και απλά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθουν το, το, ε, το αντίθετο. Δεσμεύουμε τα χρήματα και τα οριοθετούμε. Ε, τους λέμε είναι ελεύθερη επιλογή, αλλά μεταξύ αυτών των συγκεκριμένων. Όχι, να είναι συγκεντρωμένη προσπάθεια, εντάξει, αλλά όχι τόσο περιοριστική. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι ευθύνη των περιφερειών η συγκέντρωση ή μήπως των κρατών μελών. Πάντως όχι δική μας από τον κανονισμό, τον κεντρικό που να κλείνει κάθε άλλη δυνατότητα και να την αποκλεί. Ευχαριστώ. Σαλβατόρε Καρόνα. Πάρα πολύ σύντομα. Να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω, όπως έλεγε και η Κώσταν Σκρέλ, ένα θέμα το οποίο δεν ήταν δεδομένο. Δηλαδή ένας, μια συμφωνία, αν θέλετε, ανάμεσα στις προτάσεις τις οποίες κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών και στις προτάσεις τις οποίες συζητάμε εμείς στην Επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν ο τελικός στόχος του να έχουμε δηλαδή μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για τις περιφέρειες αλλά και εμείς να έχουμε μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο είναι κάτι το οποίο θα το πετύχουμε ευκολότερα. Οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και για την απλοποίηση και για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησής μας. Και γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία να καταστήσουμε την σχέση αυτή με την Επιτροπή των Περιφερειών ισχυρότερη. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω συνοπτικά θα παρουσιάσω γιατί το θεωρώ σημαντικό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. θα είναι, ποιο θα είναι το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια απορία την οποία θα χαρακτήριζα αποφασιστικού τύπου. και σε σχέση με τις λεγόμενες υπομετάβαση περιφέρειες, περιφέρειες σε μεταβατική φάση, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις στα πλαίσια της Επιτροπής μας σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργία αυτής της κατηγορίας δεν είναι κάτι το κακό, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει ή να τιμωρεί με κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες κατηγορίες. Συνεπώς η οικονομική διάσταση παίζει εδώ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να ξέρουμε τι πιστώσεις θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας υπενθύμησε η Κώσταν Σκρέλ θεμα το οποιο μας υπενθυμησε η κωσταν Σκραλ αφορα την λεγόμενη πραγματικότητα των αστικών περιοχών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα εξετάζουμε με το ίδιο ενδιαφέρον εμείς και η Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ προσωπικά εδώ θεωρώ ότι πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στη σχέση την οποία έχουμε με την Επιτροπή των Περιφερειών για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τα μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας και να κάνουμε πραγματικότητα μια καινοτομία θα έλεγα την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το να υπάρξει δηλαδή στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής μια ειδική δράση για τις περιφέρειες των πόλεων. Τι σημαίνει αυτό τώρα για ένα κράτος μέλος, τι σημαίνει αυτό για μια περιφέρεια. Αν εκ των προτέρων δεν έχει υπάρξει μια πιο εκλεπτισμένη επεξεργασία των αναγκών και των δυνατοτήτων, εάν δεν έχει υπάρξει ακόμα η σωστή επιλογή των αστικών περιοχών, των πόλεων να το πω πιο απλά, που θα ωφεληθούν, εδώ έχουμε ένα θέμα. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στην περίπτωση αυτή των ε, περιοχών ε, γύρω από τις αστικές συγκεντρώσεις. Ευχαριστώ Ερίκα Μάνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την κυρία ε, Μπρέσο και τον εισηγητή μας ε, για τα όσα μας παρουσίασε. Θα είπε και η το θέμα των πόλεων και ιδιαίτερα τη διασταυρωμένη χρηματοδότηση. Για μένα η αστική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική Μέχρι τώρα αυτά που γίνονται είναι καλά, εντάξει, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι τα μέσα και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματικά θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά αυτή την πλατφόρμα των πόλεων, συμφωνώ με τον εισηγητή. Δεν θέλω να αρχίσουμε τώρα να δημιουργούμε τέτοιες δραστηριότητες που να επικαλύπτει μία την άλλη. Και τι είναι αυτή η ιστορία με το κατάλογο των 300 πόλεων. Δεν έχω καταλάβει. Ποιε πόλει θα ενταχθούν εκεί και ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ποιο τι διαλέγει. Δεν είναι καθόλου σαφές για μένα. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς 300 πόλει με βάση κάποια κριτήρια τελείως ασαφή και συγκεκριμένα. Και μετά, από χώρα σε χώρα, διαφέρουν οι πόλεις, οι υποδομές τους, έχουν διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές προκλήσεις. Και άλλο είναι μια πόλη σε μια περιφέρεια στη χώρα μου, τη Φινλανδία, δεν έχουμε μεγάλες πρωτεύουσες περιφερειών. Ενώ αλλού στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλοι κόμβοι, μεγάλες περιφερειακές πόλεις που είναι ε, σημαντικές για την ευρύτερη περιφέρεια. Δεν μου αρέσει αυτός ο κατάλογος, δεν είναι αρκετά σαφής, ούτε δίνει ακριβή εικόνα. Κάτι άλλο που είπε ο Γιάννο Όλμπριχτ και συμφωνώ μαζί του είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ευελιξία. Ακριβώς, αυτό χρειάζεται. Και τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν εκείνα για το περίφημο 5%. Πώς θα το διαθέσουν, πώς θα το κατανείμουν στις πόλεις και από εκεί και πέρα εκείνες στα διάφορα προγράμματα και έργα τους υπάρχουν θέματα όπως είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα. και βεβαίως χρειάζεται ευελιξία και θα βοηθήσει πάρα πολύ και την αστική ανάπτυξη. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Για τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση συμφωνώ με τον εισηγητή και ελπίζω να ευδοκιμήσει η πρότασή του. Τώρα, έχω μια ερώτηση να του κάνω. για τον κανονισμό. Θα ήθελα να μάθω, κύριε Όλμπριχτεν, υπάρχει η δυνατότητα με τον κανονισμό να υπάρξει διασταυρούμενη χρηματοδότηση, γιατί δεν το λέει αυτό ρητά. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ματσόνη. Με την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών νομίζω ότι έχουμε ένα σημείο αναφοράς πλέον για την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουμε σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών στην ουσία ενισχύει τα σημεία τα οποία εμείς οφείλουμε να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο και ο καθένας από εμά θα πρέπει να ελέγξει τις τροπολογίες τις οποίες σήμερα ίσως έχουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα να εξετάσουμε προσεκτικά. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να διανύσουμε θα έλεγα ένα χρήσιμο διάστημα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε σωστές θέσεις. Καταρχάς συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που μίλησαν πριν από μένα. Είμαι πολύ συνοπτική γιατί δεν υπάρχει χρόνο σχετικά με τις εταιρικές αυτές συμβάσεις. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι εταίροι οι οποίοι προσυπογράφουν τις συμβάσεις αυτές και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη στιγμή αν θέλετε τη συμμετοχή, τη συναπόφαση, η οποία θα εμπλέκει και την κοινωνία των πολιτών με τη νομική προσυπογραφή σε εισαγωγικά, τη δεσμευτική στιγμή δηλαδή έναρξης της ισχύω της σύμβασης. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε πόσο δεσμευτικές είναι οι συμβάσεις αυτές και ποιες είναι οι πιθανές συμβάσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων που προϋποθέτει. Για την θεματολογική στόχευση ή συγκέντρωση αν θέλετε. Το κείμενο εργασίας νομίζω ότι θα μας δώσει αρκετή τους σωστούς προσανατολισμούς. Έχει σημασία να εμείνουμε σε αυτή τη συγκέντρωση των στόχων, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά τις δυνάμεις που έχουμε και ταυτόχρονα θα αποκτήσουμε και μια μεγαλύτερη ευελιξία εφόσον ξεπεράσουμε και τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί νομίζω ότι αυτά θα τα αποφασίσουν οι περιφέρειες οι ίδιες μέσω του σωστού εντοπισμού των χαρακτηριστικών και των αναγκών κάθε περιοχής σχετικά τώρα με την αρχή της αιρεσιμότητας. Έχω την εντύπωση ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο μας είπε η πρόεδρος Μπρέσο για την απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αγκυρώσει την πολιτική συνοχή στην μακροοικονομική λεγόμενη πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα αναφλέξει ε, τα πράγματα ε, και θα επηρεάσει αρνητικά τους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής αυτή η στρατηγική επιλογή βρίσκεται εν πλήρη αντιθέση με τους, στόχου στόχους της ίδιας της πολιτικής συνοχής. Σχετικά τώρα με τα μέτρα και την πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πόλεων. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Άλμπρεχτ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε οι ορισμοί αυτή οι ποσοτική η οποία περιορίζεται στο λεγόμενο 5%, να αντιπροσωπεύει μεν ένα ελάχιστο το οποίο δεν μπορεί να την χάνει παρεκκλήσεων, όχι όμως σε επίπεδο ποσοτικό. Γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ε, θα απομακρύνουμε την ποσοτική προσπάθεια ορισμού και θα στοχεύσουμε σε μια μεγαλύτερη όσμωση ανάμεσα στα, δύο, στα τρία μάλλον τα μία, κάτι το οποίο θα δώσει πολύ περισσότερο χώρο δράσης στους τοπικούς πρωταγωνιστές, σε αυτούς οι οποίοι πρέπει, αυτούς οι οποίοι πρέπει να ορίσουν σωστά την αρχή του προγραμματισμού και του σχεδιασμού. Πάντα για τις πόλεις, τις αστικές περιοχές Υπογραμμίζουμε εδώ πώς οι επενδύσεις ε, ε, οι οποίες είναι απαραίτητες για να, τεθούν σε, να τεθούν σε εφαρμογή ε, τα προγράμματα για τις περιφέρειες δεν θα πρέπει να βλάπτουν το σύνολο, το, το υπόλοιπο των περιφερειών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα μόνο για την ανάπτυξη ίσως των πόλεων, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την χωροτακτική ανάπτυξη η οποία βασίζεται ίσως στις πόλεις αλλά δεν αγνοεί τις υπόλοιπες περιφέρειες γύρω από τις πόλεις και τις υπόλοιπες περιφέρειες και την Ήπεθρο και τις παράκτιες περιοχές ανάλογα με τη χώρα. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστό σχεδιασμό και να χρησιμοποιήσουμε σωστά την χρηματοδότηση την οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ο Γιάνν Όλμπριχτ στα σύντομα. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο και να διευκρινίσω ορισμένα στοιχεία. Καταρχήν, σχετικά προς την συνάδελφό μας. Δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει κατάλογος των βασικών 300 ε, πόλεων. Ήταν μία πρόταση η οποία ήταν συνδεδεμένη με το 5%. Ε, αυτός ήταν ο κατάλογος από τη μια μεριά για την πλατφόρμα και από την άλλη πλευρά για, τον, για το πρόγραμμα. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργήσουμε ε, και στην πλατφόρμα και στις συμφωνίες συνεργασίας αυτό το κατάλογο. Η συζήτηση αυτή τώρα είναι παροχημένη διότι δεν υπάρχει τέτοια, τέτοιος κατάλογος σχετικά με το 5% πρέπει να θυμόμαστε και να έχουμε συνείδηση ότι σε πολλά κράτη-μέλη αυτό που νομίζουν ότι θα υπάρξει 5% ε, για τις πόλεις δεν είναι σωστό. Για τις πόλεις ε, θα υπάρχει χρηματοδότηση χωρίς όριο. Αυτά είναι ε, για τα συνεχιζόμενα προγράμματα παραδείγματος χάρη για τις ε, λειτουργικές ενδοχώρες των πόλεων διότι ε, τα, ε, τα η χρηματοδότηση αυτή δεν καλύπτει μόνο τις ε, πόλεις αλλά και την περιφερειά τους και ε, τελικά αναφέρθηκα στην, στην θεματική συγκέντρωση η οποία επίσης είναι ανεξάρτηση από το 5% είναι οριζόντια, είναι ένα διαφορετικό στοιχείο και ε, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταργήσουμε. Δεν είναι κανείς στο κατάλογο αυτό, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Ε, Λομπέρ. Περίμενα να μιλήσω και καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε μια πιο πλούσια ανταλλαγή απόψεων με τους παρισταμένους και ε, την πλήρη ε, εμπλοκή της Επιτροπής Περιφερειών. Εγώ, μένα λοιπόν, η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι η Επιτροπή Περιφερειών επί χρόνια έχει ε, τοποθετηθεί και προσπαθεί να διευκρινίσει την θέση της, των πόλεων στην περιφέρεια και στη συνοχή και έτσι μπορούμε να διευκρινίσουμε τις έννοιες όπως η επικουρικότητα, η αρχή της συνεργασίας, η συγκεκριμένη προσέγγιση που αναφέρεται ή στην παραγωγή και ούτω καθεξής. Προετών λοιπόν είχαμε δει ότι η Επιτροπή Περιφερειών προέβη σε έναν έλεγχο ε, της πρακτικής και στην αρχική, στο αρχικό πρόγραμμα και τώρα στην Ατζέντα 2020. Και βλέπουμε τώρα και είναι πολύ λυπηρό ότι πολλές χώρες δεν υιοθέτησαν τις ε, προτάσεις ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πόλεων. Σαν εισηγητής λοιπόν είμαι σε μια δυσχερή θέση διότι πρέπει να δώσω ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το οποίο ε, μας απασχολεί σήμερα δηλαδή την αρχή της συνεργασίας και αυτό το μέσον διότι θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δούμε πώς θα την προσεγγίσουμε. Γιατί λοιπόν να μην την αναστρέψουμε και να πούμε ότι θα καταρτιστεί από κάτω προς τα πάνω και αν το κράτος δεν συμφωνήσει με ό,τι ε, καταρτήσαμε ας το συζητήσουμε αλλά προς το παρόν πρέπει να συμφωνήσουμε θα ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω για την κατάρτιση αυτού του κειμένου και δεύτερον, εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι όλα τα κράτη θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Ε, και υπήρχε το ε, εδαφικό σύμφωνο σε ορισμένες περιοχές. Υπάρχει λοιπόν μια νέα κατάσταση, μηδενική. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι ε, εταίροι, πώς συνεργάζονται, πώς εργαζόμαστε σε αυτό το κράτος. Είναι υπεύθυνο το Υπουργείο, μετά το Υπουργείο διαβουλεύεται με την περιφέρεια για να καταρτιστεί το Εθνικό Σύμφωνο Συνεργασίας και που θα περάσει από το Κοινοβούλιο ή τέλος πάντων ποιες είναι οι αρχές, σε ποια κράτη που εμπλέκονται. Ο Γιάνν πολύ σωστά είπε η κατάσταση αλλάζει από το ένα κράτος στο άλλο οπότε πρέπει να δεχθούμε την διαφορά την πολιτιστική η οποία δέχεται να υπάρχει στις διαπραγματεύσεις στη συνέχεια το Συμβούλιο ίσως προσπαθήσει να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο αυτό το κείμενο. Αν έχουμε λοιπόν ε, ιδέες θα τις συζητήσουμε με τον Λουκ Βαντεμπράντε που ήταν ε, ε, στην Επιτροπή Περιφερειών και είναι τώρα σύμβολος του κυρίου Χάν στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο για να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το κείμενό μας γιατί σε περίοδο κρίσεως ενδεχομένως μπορεί να είναι τόσο άσχημη κατάσταση στα δημοσιονομικά μιας χώρας ώστε το κράτος αυτό να προσπαθήσει να καλύψει τα πάντα από τον προπολογισμό συνοχής σε κρατικό επίπεδο. Και αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται κάθε μέρα. Μετά, η αρχιτεκτονική της πολιτικής. Υπάρχει η ε, επιστολή των εννέα κρατών, οι οποίες είπαν ότι ε, σέβονται την, ε, το πρόγραμμα συνοχής για τις φτωχότερες περιφέρειες και ουσιαστικά ξεχνούν ότι το, η πολιτική συνοχής πευθύνεται στο μέλλον. Θέλει να προσαρμοστεί στο στόχο της Ευρώπης του 2020, πράγμα το οποίο έχει ξεχαστεί, ε, έχει παραμεληθεί. Δεν βλέπουμε να υπάρχει εδώ ένα δημοσιονομικό μέτρο για την Ευρώπη του 2020 και η συνοχή είναι και φορέας της πολιτικής και της ε, παραδοσιακής και της σύγχρονης αλλά είναι και ένας από τους στόχους ε, της πολιτικής του 2020 χωρίς όμως να καλύπτεται από χρηματοδότηση πρέπει να το δούμε και αυτό, διότι πρέπει να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια στη συνεργασία με το Συμβούλιο, διότι το κράτος είναι αυτό το οποίο αποφάσισε να προωθήσει την ε, Ευρώπη του 2020 και τώρα δεν μπορούν να μας πούνε ότι κάνουμε πίσω και δεν ε, συμμετέχουμε σε αυτό τον ολοκληρωμένο προϋπολογισμό που θα χρειαστεί συνοχή τα επόμενα χρόνια. Ήθελα λοιπόν να πω μερικά λόγια που αναφέρονται στις αρχές και όχι μόνο στις τροπολογίες. Χαιρόμαστε που είστε τώρα εδώ, διότι η Κωνσταντσα και εγώ οι συγητές των ε, διαφόρων ε, πολιτικών ομάδων μπορούν να διατυπώσουν τροπολογίες. Έχουμε ήδη προετοιμάσει ορισμένες ιστοσελίδες σχετικά με τα βασικά θέματα που έχουμε στο έγγραφο. Έχουμε εδώ 11 σημεία και ε, έχουμε σε αυτό το επίπεδο τις τροπολογίες. Δεν έχουν συζητηθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά θέματα μπορούν να γίνουν αργότερα. Αλλά τώρα αυτό που έχει σημασία είναι να διαγράψουμε τα βασικά σημεία που τονίζει στην ε, γνωμοδότησή του η Επιτροπή Περιφερειών να ε, καταρτήσουμε την έκθεση, να την έχουμε έτοιμη για τις 8 Μαΐου και αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Για αν έχεις τις ιδέες σου για τις πόλεις όπως είπε και η Κωνσταντσα, ίσως ε, είναι κάτι καινοτόμο το οποίο χρειαζόμαστε διότι δεν έχουμε αντιληφθεί τι θα γίνει αν υπάρχει μια νέα πλατφόρμα, τι θα γίνει στη χώρα, πώς πρέπει να προχωρήσουμε στη δικιά μου χώρα, στο Λουξεμβούργο ή τέλο πάντων σε κάποια άλλη. Έχουμε μια ευθύνη ότι αυτή η γενική ομπρέλα που καλύπτει τις οργανώσεις είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ε, ε, ένας πυρήνας και ε, υπάρχουν και οι μεγάλες πόλεις. Είναι βασικά θέματα τα οποία μας ενημερώνουν στα πλαίσια αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης δεν είναι κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Συμφωνώ ότι μας βοηθά, βοηθά και μας και εσάς για να διατυπώσουμε τροπολογίες και να τις ετοιμάσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Ε, όχι με τον, ε, δεν ήμουν στον κατάλογο αλλά μίλησα. Ευχαριστώ. Θέλω να αφήσω όμως ε, την Κωνσταντσα μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Μερσέντες Μπρεσό θα είναι η τελευταία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Ε, ευχαριστήσω μόνο για τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα και δείχνει ότι αυτά τα σημεία που συζητήσαμε σήμερα μας βρίσκουν πολύ κοντά στις απόψεις μας και θα μας βοηθήσει για τις αποφάσεις που επίκυνται. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πραγματικά, Πρόεδρε, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μιλήσει και για αυτό το θέμα ε, την ε, χρηματοδότηση από πολλά ταμεία σε επίπεδο έργου, γιατί αυτό θα ήταν πραγματικά επαναστατικό και χρήσιμο να έκανε αντίστοιχη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ε, Νικόλας Μάρτιν, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι ενώπιό σας για την περαιτέρω συζήτηση για τον ε, κοινό κανονισμό και την ευκαιρία που μου δίνετε να ακούσω την παρουσίαση της κυρίας Πρέσο ε, της Επιτροπής Περιφερειών για τη δική της γνωμοδότηση. Πολύ σύντομα θα ήθελα να επανέλθω στα τρία βασικά σημεία που συζητήθηκαν. Το θέμα των πόλεων, το θέμα της απλοποίησης και ε, η διασταυρούμενη χρηματοδότηση, τα πολλαπλά ταμεία και ιδιαίτερα να επανέλθω σε αυτό το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της συμβάσης εταιρικής σχέσης που προηγουμένως ανέφερε και η κυρία Μπρέσο, αλλά και άλλοι. Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το θέμα των πόλεων. Ξεκάθαρα εξήγησε το σκεπτικό της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Όλμπριχτ με τρόπο πάρα πολύ σαφή. Δεν πρόκειται για τις επεθύσεις στις αστικές περιοχές που ξεπερνούν το 5%. Ξέρουμε, κάθε είδους επενδύσεις ε, γίνονται σε αστικές περιοχές, υποστήριξη της συγκοινωνίας, της αηφορίας των μικρομεσαίων. Εδώ το σκεπτικό είναι να δώσουμε ένα ιδιαίτερο ρόλο στις πόλεις στη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης των προγραμμάτων. Και ε, ψάχνουμε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρούμε κάτι που να δρομολογεί αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό προτείνουμε το 5% ως κατόφλι ελάχιστο ε, που να συνδέεται με τις ε, ενοποιημένες ολοκληρωμένες δράσεις. Είναι ένας καταλήτης για να συμμετέχουν οι πόλεις στις δράσεις αυτές και να έχουν ένα πραγματικό ουσιαστικό ε, λόγο και στη χάραξη των προγραμμάτων αλλά και στην υλοποίησή τους. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και αυτό κρύβεται πίσω από το σκεπτικό που μας οδήγησε σε αυτή την πρόταση. σε ό,τι αφορά αυτές τις λειτουργικές αστικές περιοχές. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εμεί δεν αποκλείουμε κανέναν ε, το πεδίο εφαρμογή να είναι μεγαλύτερο και να επεκτείνεται κι αλλού, αλλά δεν θέλουμε εμείς να υπαγορεύουμε ε, ποια περιοχή είναι αυτή. Θέλουμε να αφήσουμε ελεύθερη επιλογή, ευρύτερη στα κράτη-μέλη. Ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών και το κατανοούμε. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ πιο στοχευμένο, ακόμα και σε μια ιδιαίτερη ε, περιοχή της, της πόλης, ε, συνοικία. Ή σε άλλες περιπτώσεις είναι ολόκληρη η πόλη, ενώ ε, σε κάποιες άλλες μια ευρύτερη αστική περιοχή. θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σχεδιασμού ή διατύπωση στρατηγικής μας. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση. Η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση. Η γενική χρηματοδότηση, Global Grant, ε, είναι άλλο μέσο, είναι άλλος τρόπος ε, να δοθούν επενδύσεις είναι αντίστοιχο με την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση μεν, αλλά δεν έχει την ίδια ευελιξία. Γιατί το σύνολο της διαχείρισης και της εφαρμογής πηγαίνει σε ένα διάμεσο φορέα και ε, βλέπουμε από τις απαντήσεις των κρατόμελων ότι διστάζουν να αναθέσουν τα πάντα σε πόλεις που να μην έχουν την πλήρη διοικητική δυνατότητα. Και το μοντέλο ITI της ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης ας πούμε της στρατηγικής, της ε, χάραξης, της επιλογής του προγράμματος, αλλά όχι κατά ανάγκη και τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης, τον οικονομικό έλεγχο. Αυτό μπορεί να το κρατάει η διαχειριστική αρχή. Ενώ όταν είναι συνο... λογική ε, γενική χρηματοδότηση Global Grant θα πρέπει να είναι ο ίδιος φορέας που αναλαμβάνει τα πάντα. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο τώρα και την πλατφόρμα των πόλεων. Νομίζω έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση για τον κατάλογο των πόλεων που θα συνεισφέρουν στο 5%. Είχαμε σκεφτεί να καταρτιστεί ένας ενδεικτικός κατάλογος πόλων. Ακούσαμε πολλά από τα κράτη-μέλη και καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται πραγματικά ένας κατάλογος, αλλά ένας τρόπος επιλογής των κρατών μελών τις αρχές, τα κριτήρια, τη μέθοδο, όχι ένα προκαθαρισμένο κατάλογο. Γιατί κατανοούμε ότι μπορεί να είναι πολύ νωρί για ένα κράτο μέλος να έχει ορίσει, να έχει καταλήξει σε όλε τι πόλει που μπορούν να επωφελούνται από αυτέ τι δράσει και να τι αναλαμβάνουν. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, είμαστε πρόθυμοι να προσαρμόσουμε, να ξανακοιτάξουμε το κείμενο. Ο δεύτερο κατάλογο που αναφέρεται εδώ είναι η πλατφόρμα για την ανάπτυξη των πόλεων. Γιατί υπάρχει τέτοια πλατφόρμα, και γιατί δεν είναι επικάλυψη. Διότι είναι πάρα πολύ στοχευμένη. Τι σκοπό έχει να εξασφαλίσει. Αυτό το 5% της ολοκληρωμένης δράσης για την ανάπτυξη ε, της πόλης να είναι επιτυχία. Το συνδέουμε με τις ε, καινοτόμες δράσεις στις αστικές περιοχές που θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα 0,2% που έχει Έχει προσημειωθεί. Συνδέονται λοιπόν αυτές οι δύο δράσεις και πραγματικά υπάρχει χώρος χωρίς επικάλυψη για ένα πολύ στοχευμένο μηχανισμό που να συνδέεται τα δύο. Αλλά και πάλι εδώ είμαστε πρόθυμοι να ε, κοιτάξουμε ποιος θα συμμετέχει στην πλατφόρμα αυτή. Στην αρχή η πρόταση βασιζόταν στο ότι θα ήταν καλύτερο να είναι μικρός ο αριθμός των πόλεων περιορισμένος. Στην πράξη όμως αυτό προκαλεί δυσκολίες στη διαδικασία επιλογής. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πρόθυμη να το ξανακοιτάξει, να το προσαρμόσει για να μπορούν όλες οι πόλεις να υποφελούνται αυτόματα εκείνες που λαμβάνουν το 5% μαζί με τις υπόλοιπες που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις. Διότι έτσι ε, φτάνουμε στο στόχο μας. Νομίζω αυτό θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το διευρυνήσουμε στις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με τον αρμόδιο συγητή. Έρχομαι τώρα στη διασταυρούμενη βρούμε χρηματοδότηση. σε αυτή τη διασταυρώμενη χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει στις προτάσεις της την δυνατότητα μια στήριξη ενός προγράμματος από διαφορετικές πηγές. Άρθρο 55 παράγραφος 8 λέμε συγκεκριμένα ότι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να λάβει στήριξη οικονομική από διαφορετικέ πηγέ, από διαφορετικά ταμεία. Έχετε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό συνδέεται ε, ακριβώς και με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ταμεία και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ESF. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτούς τους λόγους δεν θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί η διασταυρωμένη χρηματοδότηση. Θεωρεί ότι μπορεί και να μειωθεί κιόλα γιατί είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τα κράτη-μέλη και είναι ταυτόχρονα και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο στη χρήση πρέπει κανείς να εφαρμόζει δύο σύνολα κανόνων για την εξέλιξη θα έλεγα μίας, ενός προγράμματος. Ένα με το περιφερειακό σαν παράδειγμα ταμείο και από την άλλη ένα με το ε, κοινωνικό ταμείο. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε δίνει κάποιες δυνατότητες απλοποιώντας τα πράγματα. σχετικά με το θέμα της απλοποίησης. Εδώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι αυτό το οποίο κάνουμε με τις προτάσεις της Επιτροπής είναι να απλουστεύσουμε τη ζωή τη δική μας. Το αναγνωρίζουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή που είναι υπεύθυνη σαν παράδειγμα για τους ανθρώπινους πόρους, βλέπουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας αν μειώνονται συνεχώς οι πιστώσεις οι διαθέσιμες τα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι προτάσεις για λειτουργίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όλο και περισσότερο απαιτητικά. Βλέπετε επίσης και στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση και στην προσούρα την οποία έχει εκδώσει στον τομέα της συνοχής. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα το λεγόμενο e-cohesion είναι ένας καλός τρόπος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιες μορφές απλούστευσης. Εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα ήταν θετικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα έχει πει ότι ε, υπάρχουν πλέον οι τεχνικές προδιαγραφές, συνδέονται και είναι συμβατές με τη λεγόμενη τεχνική ε, ηλεκτρονική ημερήσια διάταξη και ταυτόχρονα είναι δυνατόν να υπάρξει ένα πόρταλ ανοιχτής, ανοιχτού λογισμικού για τις διάφορες χώρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπου αυτό είναι απαραίτητο σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Νομίζω ότι έχουμε ένα επιπλέον κλειδί για να διευκολύνουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Τέλος, για το θέμα της πολυεπίπεδης ε, διαχείρισης και της συμβάσης. Αυτό το οποίο λείπει από τις προτάσεις τις οποίες κάναμε είναι ο λεγόμενος κώδικας συμπεριφοράς. Όπως ακριβώς κάναμε προηγουμένως ε, και για το κείμενο εργασίας για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες με ένα αντίστοιχο έγγραφο με στοιχεία τα οποία θα συναποτελούν αυτό που ονομάζεται κώδικα συμπεριφοράς. Αυτό το οποίο θα λέμε είναι ότι πράγματι υποστηρίζουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στον ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και τον ρόλο τον οποίο θα παίξουν οι υπόλοιποι εταίροι. Αναγνωρίζουμε επίση σε ορισμένε ότι σε ορισμένες περιπτώσει οι περιφερειακέ αρχέ είναι οι διαχειριστέ, είναι οι βασικοί παίκτες και στη σχεδίαση και στη διαχείριση του προγράμματο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί ακριβώς στα πλαίσια του εγγράφου που θα δημοσιεύσουμε. Για τον τρόπο με τον οποίο τώρα η σύμβαση θα συγγραφεί, θα διατυπωθεί. Όπως ήδη έχουμε ε, ξεκαθαρίσει, θα ξεκινήσουμε από την αναγνώριση της ε, ποικιλία η οποία θα χαρακτηρίζει την ε, σύμβαση, τις συμβάσεις αυτές. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός αποκλειστικός τρόπος που να ταιριάζει σε όλους. Θα υπάρχουν βέβαια κάποια ελάχιστα βασικά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά θα υπάρξει και αποδοχή του ότι σε ορισμένες χώρες θα είναι εκ των κάτω προς τα άνω και σε άλλες το αντίθετο ή λιγότερο από ότι ε, σε άλλες. Λοιπόν, ε, αυτά μένει να διευκρινιστούν σχετικά με το εδαφικό πακέτο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εντάξουν τα κράτη-μέλη στα προγράμματά τους, αλλά σε, ορισμένες, σε χώρες μέλη κάτι τέτοιο δεν θα τύχει ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Αλλά εδώ τουλάχιστον ο κώδικας συμπεριφοράς θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά κάποια ελάχιστα επίπεδα για τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις αποφάσεις τις οποίες θα καταλήξουμε. Θυμίζω ότι οι μηχανισμοί λειτουργικοί παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω βέβαια ότι και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών θα παρακολουθούν το τι ακριβώς κάνουν τα κράτη-μέλη μέσω ακριβώς αυτών των μηχανισμών διακυβέρνησης. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Εάν είχαμε τους ίδιους ε, κανόνες ε, για την ε, πολλαπλή χρηματοδότηση θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε πολύ περισσότερα. Πρέπει όμως να σεβαστούμε ορισμένους κανόνες και αν δείτε τους κανόνες του βασικότερου ταμείου που εμπλέκεται σε αυτή την χρηματοδότηση θα το δούμε από εδώ. Η κυρία Μπρεσό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερους τους εισηγητές, ε, όχι μόνο για την αξιολόγηση, αλλά για, για τις πολλές ερωτήσεις τις οποίες διατύπωσαν. Επειδή είναι ακριβώς τόσες πολλές, δεν θα μπορέσω προφανώς να επέμβω σε όλα τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι στη συνέχεια θα υπάρξουν ε, και οι εισηγητές στα διάφορα ταμεία, οι οποίοι θα θα επέμβουν και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Όσον αφορά το θέμα των πόλεων και της ε, πολιτικής για τις πόλεις έχουμε τον εισηγητή Όλμπριχ τον οποίον καλούμε και ε, θα εμβαθύνουμε τη συζήτηση αυτή. Αλλά εν συντομία και εμείς πιστεύουμε ότι το να υπάρξει μία πλατφόρμα ε, για τις πόλεις είναι μεγάλο κίνδυνο παρόλο ε, που εδώ μιλάμε για τις πόλεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνίες συνεργασίας. Θα, θα σήμαινε όμως κιόλας μία σταθεροποίηση των προγραμμάτων για τις πόλεις και δεν πιστεύω ότι ε, στο πρώτο στρατηγικό πρόγραμμα πρέπει να προκαθορίσουμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στις πόλεις. Θα πρέπει, γιατί έτσι ε, θα αποθαρρύνουμε και τις άλλες πόλεις από το να συμμετάσχουν σε αυτή την ανανέωση της πολιτικής για τις πόλεις που κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή το να ε, συμμετάσχουν οι πόλεις ε, θα επιτρέψει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να διαλέξουμε μερικές και να αφήσουμε στο περιθώριο ορισμένες άλλες. Πρέπει να βρεθεί ένας ε, τύπος, ε, μία μέθοδος και να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε στο επίκεντρο των σκέψεών μας την ε, πολεοδομική πολιτική και να εμπλέξουμε ιδίως ε, θέματα που επεξεργάζονται οι περιφέρειες κατά τρόπον ώστε να βοηθήσουμε τις πόλεις και να τους δώσουμε μία νέα όθηση. Ε, ένα άλλο θέμα που είναι συνδεδεμένο με αυτό είναι οι συμφωνίες συνεργασίας. Πώς εμείς τα βλέπουμε, τα, πώς εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Ε, βλέπουμε ότι σε όλα τα κράτη και ιδίως σε αυτά όπου υπάρχει ένας ομοσπονδιακός ή περιφερειακός ε, χαρακτήρας, διότι υπάρχουν ορισμένες τέτοιες ε, περιοχές όπου υπάρχει περισσότερη αποκέντρωση δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως έγινε και με τον πρόεδρο Μπαρόζο, καλούνται τα κράτη τι να να εμπλέξουν από την αρχή από την κατάρτιση της συμφωνίας στις περιφέρειες οι οποίες θα διατυπώσουν τα ε, λειτουργικά προγράμματα και ε, θα διαχειριστούν ε, τη χρηματοδότηση των πολιτικών. Και αυτό πρέπει να γίνει και για τις πόλεις εάν θέλουμε να δώσουμε μία νέα όθηση στην πολιτική των πόλεων. Θα πρέπει δηλαδή από από την αρχή οι περιφέρειες να έχουν συνυπογράψει τις συμφωνίες ε, ε, συνεργασίας και αυτό θα μπορούσε να είναι μια σημαντική όθηση και ένα κίνητρο και ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα στρέψει την προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση διότι όσο περισσότερο οι πόλεις εμπλέκονται από την αρχή στη στρατηγική αυτή η στρατηγική συγχρόνως θα μπορεί να είναι και από κάτω προς τα πάνω αλλά και συντονισμένη με το ευρωπαϊκό επίπεδο διότι διαφορετικά η στρατηγική ε, από κάτω προς τα πάνω δεν θα είναι μια ευρωπαϊκή στρατηγική και αυτό φοβόμαστε να υπάρξει είτε μία στρατηγική από πάνω προς τα κάτω ή μία διαφορετική στρατηγική από κάτω προς τα πάνω. Ενώ αν από την αρχή έχουμε συνυπογράψει τις, ε, τα προγράμματα, από την αρχή στα προγράμματα συνεργασίας θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε από κοινού λαμβάνοντας υπόψη τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη για το 2020 όλα τα κίνητρα μέτρα. Υπάρχουν η Ευρώπη για το 2020, τα κίνητρα για τις πόλεις, τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Δηλαδή υπάρχει μία πληθώρα με και επικάλυψη προγραμμάτων που δεν επιτρέπουν να μπορέσει να γίνει σωστός προγραμματισμός αποκεντρωμένος, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της περιφέρειας ε, και ε, κρατώντας τον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει δηλαδή να υιοθετήσει καταρχήν η περιφέρεια αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να συμμετάσχει ενεργά. Είναι προφανές ότι στη συνέχεια και αυτό το είδαμε και το είπαμε πολλές φορές ότι θα υπάρξουν ε, και διαφορές αναλόγως με τη δομή του κράτους. Στα ομοσπονδιακά κράτη η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή όλων των παραγόντων από την αρχή. Όσον αφορά τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές που ανέφερε ο κύριος Όλμπριχτ, εμείς ε, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με αυτές τις στρατηγικές. Είναι πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρον εγχείρημα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και ένας τρόπος να επιτύχουμε εδαφική συνοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η πολιτική για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές διευκολύνοντας και την διεθνική χρήση των πόρων διότι ότι γιατί καταρτήσαμε αυτές τις στρατηγικές, τι ε, επιδιώκουν όλοι αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις ε, ε, μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν, να συνυπολογιστούν και έρχομαι τώρα στο θέμα της απλοποίησεως και των λύσεων που θα απορρεύσουν από την συνοχή ε, και την, ε, το ε, συντονισμό των ψηφιακών συστημάτων. Προσέξτε όμως, η απλοποίηση θα πρέπει να ακολουθήσει και την πληροφορική, διότι διαφορετικά θα βρεθείτε μπροστά σε έναν τοίχο. Αυτό έχει γίνει σε πολλούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν πληροφορική και δεν μπορούν να διέλθουν από το τείχος προς μόνο και ενός λογισμικού το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου και στο σκεπτικό σου. Για να υπάρξει λοιπόν απλοποίηση δεν θα χρειαστεί μόνο να υπάρχει μεγαλύτερη απλοποίηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σομίας Γενικεύσεως των Πολιτικών και των Διαδικασιών διότι η διαφορά διαφορετικές διαφορές στην Ευρώπη αυξάνονται συνέχεια και η πραγματική επικουρικότητα είναι το να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις πολιτικές και τους στόχους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουμε προσαρμόζοντας την στην πραγματικότητα της περιφέρειας διότι διαφορετικά δεν θα επαναφέρουμε την πολιτική της Ευρώπης στην περιφερειακή διάσταση. Είναι δύσκολο να καταλάβει την πολιτική της Ευρώπης η περιφέρεια διότι είναι περίπλοκα σχήματα τα οποία περιπλέκουν οι λεπτομέρειες και οι κανόνες και ε, ε, πρέπει επίσης να εφαρμοστεί και η κοινή πολιτική, η κοινή στρατηγική. Αυτό σημαίνει επικουρικότητα. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή και αυτό το επαναλαμβάνουμε διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε τους βασικούς στόχους της της Ευρώπης στο επίπεδο της περιφέρειας και στο επίπεδο των πολιτών. Τελειώνω. Και πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική την οποία συμμερίζονται όλοι τώρα πρέπει ακόμη να εφαρμοστεί συγκεκριμένα. το τι σημαίνει ακριβώς είναι κάτι το οποίο ξεχνούμε ίσως και νομίζω ότι ε, σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά και να δούμε ποιος είναι ο λόγος των, οποί... των ρόλων που θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας σε αυτή την κοινή στρατηγική. Διότι ναι μεν έχουμε κοινέ διαδικασίες και ε, χάνουμε στη συνέχεια το κοινό αποτέλεσμα το οποίο επιζητούμε. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι βασιζόμαστε ουσιαστικά στην χρήση της απλοποιήσεως μέχρι της δυνατότητος να αποδείξουμε το αποτέλεσμα και όχι μόνο το, την τυπική εφαρμογή της διαδικασίας. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ένα κοινό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Πολλά πράγματα ακόμη βεβαίως θα μπορούσα να πω αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ε, και τρόπο και σιγά σιγά όταν θα υπάρξουν οι προτάσεις σας θα έχουμε ευκαιρία να τις συζητήσουμε πιο λεπτομερώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κλείσει η συζήτηση τώρα εδώ και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είναι η γνωμοδότηση για το κοινωνικό ταμείο το οποίο θα παρουσιάσει η Μαρία Ιριγκογιάν Περές στην Επιτροπή Απασχόλησης σκοπεύουν να κάνουν μια πιο συγκεκριμένη παρέμβαση και όχι την γενική αντιμετώπιση την οποία ακολουθούμε εμείς. Μαρία λοιπόν έχει το λόγο και σε παρακαλώ να είσαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αφού μου το ζητάτε, και για να μην επαναλάβω τα θέματα που συζητούμε για όλα τα ταμεία. Οι ανησυχίε είναι κοινέ για το κανονισμό των ταμείων. Πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε συζητήσει για το κοινωνικό ταμείο. Δεν θα επαναλάβω τη συζήτηση. Θα πω ποιε είναι οι καινοτομίε που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιστημιστική βοήθεια ε, σε σχέση με την ΚΑΠ, ε, μείωση του προϋπολογισμού, όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, δεν είναι ιδανική λύση Καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αντιμετωπιστεί. Είναι πρωταρχικό για όλους. Εξαρτάται από το πρόγραμμα αυτό ο Ευρωπαϊκός Πληθυσμός και είναι και ε, ένα ζήτημα περιφερειακής πολιτικής στην Ένωση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε ένα νέο μέσο σαν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ήθελα να σας ρωτήσω και να μου απαντήσει ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρχομαι σύντομα σε τέσσερα σημεία. Ακούσαμε και προηγουμένως ότι μειώνονται τα ποσοστά της συγκέντρωσης. Εγώ ζητώ κάτω του 10% αντί για 60, 70, 80 μπορούμε να πηγαίνουμε προοδευτικά ε, σε μείωση 40, 30 και 20 ε, περισσότερες προτεραιότητες ε, μέγιστης επένδυσης από τα προγράμματα, να περάσουμε από τα 4 στα 6 ενδεχομένω. Αυτό αφορά 20% του ελάχιστου προϋπολογισμού για την υπόθεση της καταπολέμησης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ήθελα να επιμείνω στη Σύμβαση εταιρική Σχέσης που αναφέραμε και προηγουμένως, η μετοχή των εταίρων. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει σημασία να χρηματοδοτήσουμε τη βελτίωση των δυνατοτήτων και τη τεχνική βοήθεια των κοινωνικών εταίρων των μη κερδοσκοπικών εργανώσεων για να ε, έχουν καλύτερη πρόσβαση ε, στα προγράμματα. Συμφωνώ όμω και με τον Όλμπριχτ ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια κριτήρια για την εταιρική αυτή συμφωνία. Άλλο θέμα έχει να κάνει με τον αριθμό των ε, προτεραιοτήτων και τις περιφέρειες λεγόμενες ε, με μετάβαση. Θεωρώ και εγώ ότι ε, η χρηματοδότηση περιορίζεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αλλά εγώ θεωρώ σημαντικό ότι και ε, οι περιφέρειες σε μετάβαση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και θα πρέπει να γίνουν πρόοδοι σε αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ε, μέτρα τα οποία επιδοτούνται. Θα ήθελα να ρωτήσω και σε αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μου απαντήσει. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν σημεία για να ξεκινήσει η συζήτηση για το Κοινωνικό Ταμείο, κυρία Πρόεδρε περιμένω τα σχόλιά σας και τη βοήθειά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Η κυρία Οκατσιέσκα απουσιάζει, όπως και η κυρία Μανέσκου. Η κυρία Σρέτερ παρακαλώ. Σύντομα. Να σας πω μερικά βασικά. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια εδώ και καιρό είμαστε σε καλή συνεργασία Είμαι μέλος και στην Κοινωνική Επιτροπή και σκιώδη συγγήτρια για το Κοινωνικό Ταμείο. Γνωρίζω ε, καλά σχετικά αυτό το μέσο. Υπάρχουν μερικά προβλήματα στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο είναι το άρθρο 4.3 με τον κανόνα της συγκέντρωσης. Δεν μπορεί να παραμείνει όσο έχει, πρέπει να αλλάξει απλούστατα. Και το συζητούμε αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, να επικεντρωθεί όχι στις προτεραιότητες επενδύσεων, αλλά στις θεματικές προτεραιότητες. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, είναι λάθος η προσέγγιση. Για το άρθρο 5... Ε, ποια θα είναι η πηγή χρηματοδότησης για την πολυεπίπεδη ε, διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση το άρθρο 5 ε, του Γενικού Κανονισμού και εδώ Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών και δεν έχει κανένα νόημα να γίνει κάτι τέτοιο. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να γίνεται με την ίδια ένταση σε όλες τις περιφέρειες. Δηλαδή οι εταίροι να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να είναι ενίο αυτό για όλες τις περιφέρειες. Ε, χρειάζεται αλλαγή αυτή οπωσδήποτε. Είναι μια μικρή διαγραφή, δεν είναι τίποτα. Ε, αυτά τα βασικότερα στην Κοινωνική Επιτροπή το συντελεστή στο ποσοστό είναι 20% και στο Κοινωνικό Ταμείο υπάρχουν και κάποιοι κανόνες απλοποίησης, δεν ξέρω, θα πρέπει να βελτιωθούν. Ιδιαίτερα η χρηματοδότηση ε, και τι γίνεται με το γενικό κανονισμό, γιατί έχει ειδικού κανόνες έξτρα ε, το κοινωνικό ταμείο, διαφορές από τα υπόλοιπα ταμεία. Ε, υπάρχουν και κάποια άλλα καινοτόμα και έρχομαι σε ένα ζήτημα ουσίας ε, και αρχής. Αυτό το 5% το είχαμε ένα κατόφλι για τις πόλεις. Έχει δίκιο εδώ ο Γιάννο Όρμπριχτ. Θα πρέπει να το κάνουμε για όλα τα ε, ε, μέσα και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στο Λίντερ και στην αστική ανάπτυξη, το ελάχιστο αυτό το 5% κατόφλι. Αυτά που λέει η έκθεση του Όλμπρεχτ, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα ίδια ποσοστά και για το κοινωνικό ταμείο, γιατί υπάρχει και εκεί ένα τοπικό επίπεδο, το οποίο δεν περιγράφεται αρκετά σαφώς. Για να έχουμε αυτό το τουλάχιστον 5% σε όλα τα ταμεία, σε όλα τα μέσα, με την ίδια μέθοδο. Για να υπάρχει και κάποια στοιχειώδη συνέπεια και συνέχεια εκεί για να μπορούν να συνδυάζονται καλύτερα τα ταμεία και μεθοδολογικά να είναι γνωστή, να μαθευτεί στις περιφέρειες η μέθοδος. Υπάρχει ένα άρθρο που περιγράφεται αυτό στην πράξη και ακριβώς γι' αυτό το 5% περιγράφεται η κατάσταση στο Περιφερειακό Ταμείο και χρειάζεται προσαρμογή στο κοινωνικό ταμείο για να μπορούν να αξιοποιούνται ε, στις πόλεις με την ίδια μέθοδο οι πόροι από τα δύο ταμεία. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να υπάρξει αυτή η δυνατότητα και να αλλάξει η διατύπωση, για να μπορούν ακριβώς να κουμπώνουν τα χρήματα από το ένα ταμείο στο άλλο, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιοι όροι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα και αφορούν και την εδαφική διάσταση που είναι η δική μας αρμοδιότητα εδώ στην Επιτροπή μας. Και αν περάσουν όλα αυτά νομίζω θα είναι καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Έφυγε η Κονέλια ο Ευχαριστώ να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Να συμφωνήσω με την κυρία Σέντερ, λέγοντας ότι ακόμα και αν έχουμε δύο ταμεία, ακόμα και αν έχουμε δύο επιτρόπους, θα πρέπει να έχουμε μία λογική στο σύστημα. Γιατί στο ένα ταμείο έχουμε τη θεματική συγκέντρωση και από την άλλη έχουμε τη ε, θεματική συγκέντρωση σε επίπεδο προγραμμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ θα χάσουμε το λογαριασμό. Πώς μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλά ταμεία να ακολουθούμε δύο διαφορετικές λογικές. Πώς μπορούμε να έχουμε το ITI το οποίο είναι περίπλοκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Με διαφορετικούς άξονες, με διαφορετικές δράσεις, διαφορετικά προγράμματα, γενικά ιδιαίτερα περίπλοκο. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε σαν Επιτροπή να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο σύστημα με τα ταμεία γιατί αλλιώς θα χάσουμε τον μπούσουλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Σούκοβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επανήλθατε στις βασικές αρχές για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την αλληλεγγύη δηλαδή και την κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι και η δική μας στόχη. Σε επίπεδο της συγκέντρωσης των στόχων και ανάλογα με τη συμμετοχή των περιφερειών, διαρωτώμεθα αν το να έχουμε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης μας δίνει καρπούς. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάποιες συγκεντρώσεις πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτά ορατά αποτελέσματα με ε, μεγάλα ποσά τα οποία να έχουν σαν στόχο πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. αν πούμε ότι το 40% θα το δώσουμε σε 5 ας πούμε προτεραιότητες και τα υπόλοιπα 60 σε όλα τα υπόλοιπα φοβάμαι ότι μιλάμε για πολυδιάσπαση και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για περαιτέρω συγκέντρωση του στόχου. Το EDF και το Κοινωνικό Ταμείο έχουν συγκρίσιμα επίπεδα συγκέντρωσης γιατί οι κανονισμοί λειτουργία τους είναι παρόμοιοι. Για το EFSF έχουμε 11 θεματολογικά θέματα, ενώ το Κοινωνικό Ταμείο έχει 4 ευρύτερα θέματα και 18 επιμέρους προτεραιότητες. Αυτά ανταποκρίνονται στους δικούς μας στόχους. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι προτιμότερη η συγκέντρωση να γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους και όχι σε επίπεδο λειτουργικού προγράμματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται όμως ιδιαίτερα για το Περιφερειακό Ταμείο από τα προγράμματα τα εθνικά και όχι τόσο από τα προγράμματα τα οποία εμείς υποβάλλουμε. Για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αναφέρθηκε ο κύριος Μάρτιν στην, στον, κωδικό αυτό, στον κώδικα συμπεριφοράς. Πράγματι θα πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι εταίροι από την προετοιμασία της εταιρικής σύμβασης μέχρι τη στιγμή της εφαρμογής του προγράμματος. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, να διασφαλιστεί η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών για να υπάρχει η αίσθηση θα έλεγα του ιδιόκτητου της διαδικασίας, κάτι το οποίο θα λειτουργήσει σαν κίνητρο. Η πρόταση για 5% όλων των μέσων θα πρέπει να εναλλάσσεται, αυτό είναι κάτι το καινοτόμο για μένα. μπορούμε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε εμείς πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στα πολλά επίπεδα συγκέντρωσης, αλλά αυτό είναι ίσως θεματολογικά κάτι το οποίο δεν αφορά τη δική μου γενική διεύθυνση. Τελειώσατε κυρία Σούκοβα. Η Ελίζαμπετ Μπετσέντερ. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω το θέμα της συγκεντρώσεως στο ESF. Πρέπει να σας πω όμως ότι και να το καταλάβω δεν μπορώ να το προτείνω και δεν θα δεχθώ να υπάρξει κάτι τέτοιο στο ESF διότι είναι ανόητα ε, όσον αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεις και έχω ένα πολύ καλό Παράδειγμα, υπάρχει η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Είναι από τα θέματα ε, που είναι σε ψηλές, ε, σε, στη θέση 8 ή 9 και υπάρχουν 7 προτεραιότητες. Εάν λοιπόν, ε, ε αν έχετε χρηματικά χρηματοδότηση. Θα κάνατε ε, ε, ένα πρόγραμμα για αυτό το βασικό θέμα. Θα χρειαζόσασταν όμως να έχετε ήδη και τις 7 προηγούμενες επενδύσεις για να υπάρχει νόημα στο όλο εγχείρημα. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι θα γίνει το ίδιο όπως και στο ERDF ε, όπου βασίζεστε σε τρεις θεματικές ενότητες. Γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι στόχοι και ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναφέρεται εις ε, την ε, ανάπτυξη μόνο σε ορισμένα κράτη-μέλη όπου υπάρχει καλή διοίκηση και ορισμένα κράτη το χρειάζονται ε, διότι υπάρχει μία μακρά μεταβατική περίοδος και χρειάζονται ε, υψηλή χρηματοδότηση. Όπως το ERDF λοιπόν πρέπει να βασιστεί κανείς σε τρεις θεματικές ενότητες 8, 9 και 10 ας πούμε και έχουμε 20% για την φτώχεια, αντιμετώπιση της φτώχειας. Έχουμε δηλαδή ε, τους ίδιους ε, αριθμούς, τις ίδιες συγκεντρώσεις όπως και στο ERDF και αυτό μας δίνει κάποια ευελιξία για το πώς θα επιτύχουν την, ε, τον θεματικό στόχο. Αυτό χρειαζόμαστε, την ευελιξία για να επιτύχουμε τον θεματικό στόχο. Δεν πρέπει δηλαδή να τους λέμε ότι θα γίνει μόνο με ένα τρόπο και είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Γιάννη. Δηλαδή η ίδια μέθοδος θα πρέπει να ισχύσει και στο ERDF και στο ESF, διαφορετικά το Κοινοβούλιο δεν ε, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που έχει διατυπώσει ούτε να βρει λύσεις. Ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω το λόγο στην Επιτροπή, άλλο σχόλιο. εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα σχόλια και τις απόψεις που μου είπατε. Ε, ε συμφωνώ να συμπεριλάβω με τις ανησυχίες σας για το άρθρο 4, 3 για το άρθρο 5 ε, και αυτά που μας είπε ο Άμπριθ για τη συνοχή, τη λογική συνέπεια των ταμείων. Ε, το ταμείο δεν θα πρέπει να έχει λίγο την αρχή ποτιστήρι, δηλαδή ότι δίνουμε λίγα λεφτά στα πάντα, αλλά να έχουμε μια συγκεντρωμένη και στοχευμένη και αποτελεσματική προσέγγιση. Μάλιστα, το χρονοδιάγραμμα η Πρόεδρος, μάλλον περί τα τέλη Απριλίου θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης με τις τροπολογίες και η προθεσμία θα είναι κάπου το Μάιο για την κατάθεση τροπολογιών, οπότε και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ενδεχομένως τέλη Μαΐου, όπως σας φαίνεται, ή τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Έχουμε καιρό ακόμα και για άλλα στοιχεία. Παρακαλώ σκεφτείτε από τώρα τις τροπολογίες όμως, γιατί πιέζουν οι ημερομηνίε. Ιδιαίτερα ε, οι άλλοι συνάδελφοι που είναι του Γενικού Κανονισμού φροντίστε να συνδυαστούν. Ο Βανίστεροι. Κοιτάξτε, ε, δεν πρέπει να τιμωρείται ποτέ η φιλοδοξία. Μπορεί να έχουμε προχωρήσει από τους άλλους, αλλά σε περίοδους κρίσης το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν θα πρέπει να μας τιμωρούν. Ε, σε αυτό που είπατε υπάρχει εξή αξία τώρα από πλευράς μου. Πρέπει να σας πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, η ψηφοφορία στην Επιτροπή καλώς. Ε, στην, στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή. Αλλά αν πάμε στην Ολομέλεια γιατί αυτό μας είπαν στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα στην ομάδα επαφής για τις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές και το πλαίσιο. Μας είπαν να ε, συντονίσουμε λίγο και να προγραμματίσουμε τη δράση μας, να συνδυάσουμε τα σημαντικότερα που συνδέονται μεταξύ τους. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με τους ε, εισηγητές ε, και το συζητούμε. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Αυτοί που έχουν προχωρήσει περισσότερο, τι θα κάνουμε, να τους τραβήξουμε πίσω. Εσείς είστε πρόεδρος της Επιτροπής, εσείς θα το συντονίσετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που μπορώ να τα μπλοκάρω, να τα σταματήσω και κάποια άλλα που μου διαφεύγουν. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά στη συνεδρίαση των συντονιστών. Πρέπει να τα πούμε τώρα αυτά, ο κύριος Όμπριχτ, διευκρινιστικά. μας ενημέρωσαν ότι εμείς ως εισηγητές θα πρέπει να προετοιμάσουμε το σχέδιο της έκθεσής μας, χωρίς τροπολογίες, το σχέδιο και μόνο το κείμενο που είναι τη λογική έκθεση και μετά τις τροπολογίες να είμαστε σαφείς, γιατί αν εμείς πρέπει να προετοιμάσουμε την έκθεση συν τις τροπολογίες τις συγκεκριμένες, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο έκθεσης, καταλαβαίνετε. Δεν το συζητούμε αυτό το θέμα τώρα, λέει η Πρόεδρος. Ε, πολύ συγκεκριμένα είμαστε σε ένα άλλο θέμα. Δεν είναι τη δική μα επιτροπή αυτή η έκθεση. Γνωμοδότηση κάνουμε. Και αν θέλουμε να το λάβουμε υπόψη μας, θα πρέπει να ε, προσαρμοστούμε στο χρονοδιάγραμμα εκείνη τη Επιτροπής. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που να αποφασίζονται και για τη συνοχή και για το κοινωνικό ταμείο και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το γενικό κανονισμό και πώς αυτά θα συνδεθούν. Ε, προς το παρόν δεν το ελέγχουμε εμείς, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που μας ζητηθεί. Και χρειάζεται και πολλή δουλειά. Θα τα πούμε αυτά στους συντονιστές παρακαλώ. Λοιπόν, να ολοκληρωθεί εδώ για σήμερα αυτή η συζήτηση για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Α, η Κωνσταντσα Κρέλ, συγγνώμη. Ναι. Μια μικρή παρατήρηση θέλω να κάνω για το χρονοδιάγραμμα. Δεν είχαμε αποφασίσει από κοινού με τις άλλες επιτροπές ότι δεν θα γίνει ποτέ συζήτηση, μάλλον ψηφοφορία για κανονισμό ταμείου πριν ψηφιστούν τα θέματα του γενικού κανονισμού. Να το πω αλλιώς. Εάν στους επιμέρους κανονισμούς αλλάξει κάτι που επηρεάζει και αφορά το γενικό κανονισμό, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα των επιμέρους επιτροπών. Και θυμάμαι και την Επιτροπή Απασχόλησης και ε, την απόφαση αυτή την υποβόσκουσα για το άρθρο 50. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ πέρα και δεν τα θεωρώ καθόλου συνεπή αυτά. Ναι, εγώ νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει, αλλά όπως είπε και ο Λάμπερτ υπάρχουν και άλλες φιλοδοξίες. Δηλαδή αν τελικά ε, ο γενικός κανονισμός καταλήξει αλλού, θα πρέπει να επανέλθουν οι επιμέρους επιτροπές να το ξανακοιτάξουν αυτά που ψήφισαν. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη πώς να το πω, σεβασμού της δύσκολης και πολύ δύσκολης διαπραγμάτευσης που γίνεται για το γενικό κανονισμό. Αν κάποιος δεν θέλει να το σεβαστεί θα πρέπει να υπομειστεί και τις συνέπειες. Θα το συζητήσουμε αυτό πολιτικά στους συντονιστές. Θα ήθελα να προχωρήσουμε τώρα σας παρακαλώ στο επόμενο θέμα. Είναι εδώ η Αναμυράντα. Έχουμε τρεις εκθέσεις. Δύο από τους συναδέλφους δεν είναι μαζί μας σήμερα και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους πολιτικούς συμβούλους Τεσέιρα και Βλάσεκ να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς γίνεται, πότε θα έρθουν σε εισαγωγικά τα αφεντικά σας. Και θα ήθελα να περάσουμε στο σημείο 6, γνωμοδότηση Μιράντα, για την αλληλεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή βιοτεχνική αλληλεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την προσπάθεια που έκανε και να προτείνω μια προφορική τροπολογία. Στην γαλλική διατύπωση υπάρχει ένα μεταφραστικό λάθος. Η αστρακοαλία σαν παράδειγμα στα ισπανικά υπάρχει μάλλον το πρόβλημα, υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην οστρακοκαλλιέργεια και την αλληλεία οστράκων. Στα γαλλικά η σωστή λέξη η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι conchiculture, conchiliοκαλλιέργεια. Πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για διορθώσεις διατύπωσης στα ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά. Υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις βιοτεχνικές μεθόδους και στην παραγωγή την εκτατική ε, προϊόντων οστρακοκαλλιέργειας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η παράκτη αλληλεία, η βιοτεχνική αλληλεία επηρεάζουν την οστρακοκαλλιέργεια και ε, επηρεάζουν επίσης και επηρεάζονται και από την ε, θα έλεγα εντατική ε, καλλιέργεια εκτροφής ηχθείων. Αλία η παράκτια είναι αηφόρος βιολογικά, έχει καλύπτει πάνω του 60% των εργαζομένων στον τομέα της αλίας, άμεσα και έμεσα, αλλά δεν έχουμε όμως μία σωστή θα έλεγα προσπάθεια ορισμού της παραδοσιακής αλίας και της παραδοσιακής οστρακοκαλλιέργειας. οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται έχουν ξεπεραστεί, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και οι ιδιαιτερότητες περιφερειακές, οικολογικές ε, πλευρές και επίσης να προωθήσουμε και αηφόρες μορφές καλλιέργειας. Η παραδοσιακή αλληλεία, η λεγόμενη μικρά αλληλεία, είναι η πλέον αηφόρο σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Νομίζω ότι αυτά όλα θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στον τομέα της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των παρακτήων κοινοτήτων. Αυτού του είδους ε, αλληλεία έχει επίσης και πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία, ιδιαίτερα στις ε, πλέον απόμακρες περιοχές. και αυτή η ποικιλία η πολιτισμική παίζει σημαντικό ρόλο και στην μεταφορά θα έλεγα και την διαιώνιση αυτού του είδους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν όμως και αρνητικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τις δραστηριότητες αυτές. Υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης, υπάρχουν προβλήματα μόλυνσης. Ξέρουμε τι έγινε στη Βρετάνη με το με συγκεκριμένα πετρελαιοφόρα και με τις πετρελαιοκυλίδες με το πλοίο Πρεστίζ το οποίο έφυξε ακριβώς αυτού του μορφ, αυτής της μορφής την, αλληλεία ακόμα και στη δική μου χώρα και απειλείται ακόμα και από τις, ε, από τις δραστηριότητες τις οικοδομικές στις παράκτιες περιοχές η αλληλεία αυτή. Αν θέλουμε να ορίσουμε την μικρά αυτή αλληλεία και σε επίπεδο ωφέλους κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τα επαρκή στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα στον τομέα της συνοχής. Και γι' αυτό και προτείνουμε στην γνωμοδότησή μας να συλλεχθούν ε, ε στοιχεία ε, οικονομικά και κοινωνικά με επακριβέστερο τρόπο. Πιστεύουμε επίσης ότι σε μια τέτοια εποχή κρίσης και σε μια τέτοια εποχή μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής η κατάσταση της μικράς αλληλείας όπως λέγεται εξαρτάται από τομείς ανεξάρτητους της αλληλείας. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές οικονομικές και κοινωνικο-οικονομικές λύσεις. Δεν μπορεί ένας αλλιέας που ασχολείται σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα να μετατραπεί αυτόματα σε ε, επιχειρηματία, δεν έχει τις δυνατότητες και την κατάρτιση που χρειάζεται και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση αυτής της δραστηριότητας ε, μια καλύτερη μορφή προστασία της παραδοσιακής αλληλείας και μια ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρξει στον τομέα αυτό μια πολυετή στρατηγική και στα πλαίσια της τοπικής ανάπτυξης στην οποία έχουμε αναφερθεί ήδη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε αυτήν την μικρή γνώμοδότηση η οποία όμως θα πρέπει να δείχνει το μήνυμα στήριξης πολιτικής αυτής της αηφόρου δραστηριότητας, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο τμήμα του μελλοντικού αλλιευτικού ταμείου για την αλλιευτική αυτή ε, δραστηριότητα. Να δημιουργηθεί επίσης και ένα μικρό ειδικό πρόγραμμα βοήθειας προς τη μικρά αλληλεία, ε, που θα κατευθύνεται αποκλειστικά στις ε, ε, κοινότητες της παράκτιες που εξαρτώνται από την αλληλεία έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης και να στηρίξουμε επίσης και με το πολιτικό μας μήνυμα την Επιτροπή Αλληλείας έτσι ώστε να υποστηρίξει και αυτή τη μορφή της αλλιευτικής δραστηριότητας ε, αηφόρου και σε επίπεδο ε, συνοχής. Περιμένω ε, επίσης και τα σχόλια των άλλων συναδέλφων. Από πλευρά της Γκουε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σαν σκιώδης συζητητής, λέει ο κύριος Πονγκά ευχαριστήσω ε, για τις προτάσεις και θέλω να κάνω δύο σύντομες ε, ερωτήσεις. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασκεί διάφορα είδη ε, αλληλείας και γι' αυτό δεν πρέπει να θέσουμε σε αντιπαράθεση την μικρή αλληλεία με την βιομηχανική αλληλεία διότι μπορεί και οι δύο να είναι συμπληρωματικές για την ανάπτυξη της οικονομίας μιας περιοχής. Θέλω να τονίσω την ερασιτεχνική ε, και μικρή αλληλεία στην, ε, στις παράκτιες χώρες και στις χώρες χώρες της περιφερείας της Ευρώπης. Θα διατυπώσω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και σας ευχαριστώ. Εσείς ε, είσαστε εν ονόματι του ΕΛ, κύριε Πόγκα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, ίσως ο Λαμπέρ Βαλνίστελ Ρόι. Ευχαριστώ που μου δώσατε το σχέδιό σας και το μόνο το οποίο εγώ έχω να πω από ε, τη δικιά μου σκοπιά είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει μία πολιτική αλληλείας και μάλιστα ε, η οποία να είναι η φόρος και για τα μεγαλύτερα και για τα μικρότερα ε, πλοία και ε, η χρήση ε, των δραστηριοτήτων αυτών έχει διευρυνθεί και βλέπουμε ότι τώρα στις παράκτιες περιοχές υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αυτές τις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα μπορούν να έχουν ένα εισόδημα όχι μόνο από την αλληλεία αλλά και από τον τουρισμό και από άλλες πηγές. Οπότε Θεωρώ ότι χαιρετίζουμε αυτές ε, τις ε, δραστηριότητες και μπορούν να περιληφθούν στη δραστηριότητα του ERDF, διότι πολλές φορές όταν υπάρχει ο πλήρης ανταγωνισμός από τα μεγαλύτερα πλοία δεν μπορεί κανείς ε, να προχωρήσει χωρίς τη διατύπωση μιας ουσιαστικής πολιτικής και ιδίως με το ERDF σχέση με το παρελθόν. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συναδέλφισσα, την κυρία Μιράντα, για την ε, μικρή σύντομη αυτή έκθεση. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μια ομάδα ε, αλλιών που δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, όπως είναι η παραδοσιακή μικρή αλής, που είναι κυρίως στη Μεσόγειο, που μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο θέμα της αλίας, αλλά και στο θέμα καινούριων πολιτικών για την, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, για παράδειγμα, ένα ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν και θα πρέπει να ενισχυθεί μέσα από το καινούριο Ταμείο ε, Θαλάσσιας και Αλληλευτικής πολιτική είναι η συμμετοχή του στην παρατήρηση σε σχέση με τι επιπτώσεις κλιματική αλλαγή στα θαλάσσια και παράκτα οικοστήματα. Πολλέ φορέ πριν οι επιστήμονε καταγράψουν παρόμοιε παρατηρήσει, είναι πιθανό ότι ψαράδες αυτοί παραδοσιακοί μπορούν ε, να ε, καταγράψουν τις παρατηρήσεις, όπως παράδειγμα η καταγραφή ειδών που εισβάλλουν από άλλες περιοχές λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας της θάλασσας και γενικότερα ε, της αλλαγής του κλίματος. Θα ήθελα επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πολλές φορές αυτές οι μικρές κοινότητες παράκτηνα ελαιών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές οικονομικής δραστηριότητας ε, αλλά από την άλλη μεριά έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκού επίπεδου που απαιτούν ορισμένε διαδικασίε αυστηρέ, στι οποίε δεν έχουν εύκολα δυνατότητα να ε, εξοικειωθούν. Άρα θα πρέπει να δούμε, ε, όπω αναφέρθηκε και πιο πριν, και ειδικά προγράμματα που βοηθούν αυτού πραγματικά του ε, μικρού παράκτιου ε, αλείς, με παραδοσιακό τρόπο. Και ένα τρίτο σημείο στο οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι ε, στη στρατηγική για την αποκατάσταση θαλάσσιας βιπικιλότητας, οι παράκτιες ε, κοινότητες αυτών των αλλιών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαχείριση παρόμοιων περιοχών με στόχο την ανάκαμψη της θαλάσσιας βιπικιλότητας. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όπου έχει εφαρμοστεί, σε χώρε όπου έχει εφαρμοστεί, υπάρχει πολύ σημαντική εμπειρία, θετική εμπειρία, άρα θα πρέπει να το προβλέψουμε ε, πιο έντονα στα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευχαριστώ. Thank you uh, very much. I don't see any more... Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους ομιλητές. Θέλω λοιπόν ε, να παρακαλέσω τώρα την ε, εκπρόσωπο αν θέλει να ξαναλάβει τον λόγο και μετά θα αποφασίσουμε για τις ημερομηνίε των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ευχαριστώ όλους για τις γνωμοδοτήσεις. Είμαστε ανοιχτοί αλλά δεν θέλουμε ε, να υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ της βιοτεχνικής και της βιομηχανικής αλληλείας. Είναι όπως η κατάσταση των ποσοστώσεων προς το Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει μία διαφοροποίηση κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ειδική μεταχείριση για να αποφύγουμε τις διακρίσεις σε πολλές περιπτώσεις. Στην ε, ε, βιοτεχνική Αλλοί έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αν δεν την προστατεύσουμε θα εξαφανιστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω τώρα να προτείνω σαν ημερομηνία για τις τροπολογίες 29 Μαρτίου του 12, ε, στις 12 το μεσημέρι. Και ε, κατόπιν αυτού προχωρώ στο σημείο 7 της ε, ημερησίας διατάξεως σχετικά με την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη με συντάκτη του κύριο Βλάσακ υπάρχει κάποιος άλλος ε, να μιλήσει για τον εισηγητή όχι αλλά ξεκινούν οι σκιώδεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών σχετικά με τα θέλγητρα των επενδύσεων, διότι στην περιοχή μας η κρίση έπληξε τις επενδύσεις, αλλά το 2011 σημειώσαμε μία αύξηση 5% του αριθμού των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να προσελκύσουμε επενδύσεις τα κράτη αλλά και οι περιφέρειες πρέπει να προσφέρουν συγκεκριμένα ε, προσόντα τοπικά. Αλλά τα προσόντα αυτά δεν είναι αντίστοιχα με τις ανάγκες ιδίω στην Ευρώπη και μιλάμε στην Επιτροπή Οικονομικών για ε, ε, τις οικονομικές, φορολογικές διευκολύνσεις και ούτω καθεξής. Αλλά ουσιαστικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της αλλαγής για να συμβάλλει στη σύγκληση της αναπτύξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις για την κατάρτιση δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών στα πλαίσια αυτής της συνοχής και συγχρόνως έχουμε ε, χρηματοδοτήσει ε, δύο ε, δισεκατομμύρια χιλιόμετρα δρόμων, ένα πολύ υψηλό αριθμό μικρομεσών επιχειρήσεων, διευκολύνουμε τους επενδυτές με κάθε τρόπο, αλλά για να μπορέσει αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει υπάρχει μία βασική προϋπόθεση και εδώ αναφέρομαι στις αποτελεσματικές υποδομές. Όποια επιχείρηση θέλει να επενδύσει υπολογίζει τις υπάρχουσες υποδομές. Όταν εγώ δούλευα σε μία ιδιωτική εταιρεία είχα την ευκαιρία να λάβω κάποια απόφαση σχετικά με επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι το κριτήριο αυτό της της ενδιαφέρουσας υποδομής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδρομές, όποιες και να είναι, και αυτό πρέπει να αποτελέσει μια πραγματική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω μέσω της πολιτικής συνοχής. Δεν επαρκεί όμως. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η υποδομή, χρειάζονται όμως και άλλα προσόντα των περιφερειών που θα πρέπει να προβληθούν και εδώ αναφέρουμε στην έρευνα, στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτά μάλιστα έχουν σχέση με τον σκληρό πυρήνα του θέματος, ο οποίος είναι ο εξής. Θα πρέπει οι περιφέρειες να καταλάβουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, της ερεύνης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Δεν πρέπει όμως να έχουμε μόνο μια καλή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν και σε επίπεδο των περιφερειών. Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά διακυδεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα έτη. Γι' αυτό και η υψηλού επίπεδο επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική και ιδίως εάν συνοδεύεται με την προώθηση των τεχνολογιών στις περιφέρειες. Και βεβαίως όλα αυτά σε συνδυασμό με την έξυπνη ανάπτυξη την οποία προωθεί η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Πρέπει να ενισχύσουμε και την έρευνα και την εφαρμοσμένη έρευνα και για τα νέα κρατημέλη θα πρέπει να, ε, ε, να επιμείνουμε και στην ε, εκπαιδευτική υποδομή. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η εφαρμοσμένη έρευνα, διότι αυτή τη στιγμή μόνο 2% των αποτελεσμάτων της ερεύνης εφαρμόζονται πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μόνο 2% ε, των ε, ε, διπλωμάτων μπορούν να εφαρμοστούν. Κάνουμε ε, μεγάλες προσπάθειες στον τομέα της έρευνας, προωθούμε την έρευνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, αυτές τις έρευνες ε, μέσω της παραγωγής και της βιομηχανίας και στη συνέχεια πρέπει με αυτόν τον τρόπο να υποκινήσουμε την ανάπτυξη. Είναι κάτι που τονίζω. Δηλαδή η χρηματοδότηση έρευνας δεν επαρκεί διότι έχουμε δεσμεύσει ε, ε, δισεκατομμύρια για την έρευνα δεν τα ξοδεύουμε και μεθαύριο θα βρεθούμε με αυτά τα ποσά τα οποία δεν θα έχουν διατεθεί. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η έρευνα να ε, οδηγήσει σε παραγωγή τελικών προϊόντων και τονίζω το θέμα αυτό διότι αν θέλουμε όντως να υπάρξει Ευρώπη της καινοτομίας και της έρευνας θα πρέπει πραγματικά η έρευνα αυτή να είναι παραγωγική και να μεταφραστεί ε, σε ανάπτυξη. Και γι' αυτό στο άμεσο μέλλον οι ε, περιοχές και τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να καταρτήσουν στόχους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών για να υπάρχουν προσβάσιμες διάφανες επενδύσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι ότι σε μια τέτοια κρίση και το σχετικό ταμείο είναι σημαντικό διότι υπάρχει η τάση από τους οικονομικούς παράγοντας να μειώνουν την επένδυση στον τομέα της έρευνας παραδείγματος χάρη ενώ εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αυξηθεί η επένδυση αυτή και έχουμε θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο 2-3% για τα κράτη-μέλη αλλά ουσιαστικά ε, στην πρακτική αλλάζει το θέμα αυτό. Το, τα χρήματα για την έρευνα μειώνονται ιδίω οι ιδιωτικές επενδύσεις και είναι ένα στοιχείο που πρέπει να συνυπολογιστεί διότι εντωμεταξύ ε, πρέπει να υπάρχει καινοτομία εις την ε, έρευνα. Και τέλος οι λιγότερο ανεπνιγμένες περιοχές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν επιπροσθέτως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει εδώ εδώ να έχουμε μία σαφή εικόνα της συνοχής, της αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το, την έκθεση η οποία μας απασχολεί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προβλήματα αλλά πιστεύω ότι οι τροπολογίες θα βελτιώσουν το κείμενο. Καταρχήν το σημείο 4 που αναφέρεται στα συγκριτικά οικονομικά προσόντα. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι από την άποψη αυτή μιλάμε για ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και άρα στο άρθρο 4 δεν είναι πολύ σαφής η διατύπωση και στη συνέχεια ο ε, εισηγητής αναφέρεται ή στην φορολογική πολιτική και στη φορολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες στον τομέα αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα είναι αποτελεσματική, θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να αναπτύξει αυτή την πολιτική και ελπίζω ότι η έρευνα και η καινοτομία θα βοηθήσουν και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ, πολύ. Ξενόματος του κυρίου ε, Βλάσακ, είναι ο κύριος ε, Πορέμπα νομίζω. Ναι. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει συνήθιση η διαδικασία ο κύριος Πορέμπα. Θα ήθελα να παρουσιάσω το γενικό πλαίσιο, αν θέλετε να ολοκληρώσω στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε το χρόνο που θα θέλαμε. Είναι κρίσο ο κατάλογος των ομιλητών. Παρακαλώ, όσο γίνεται πιο σύντομη να είστε. Κύριος Πορέμπα. Μάλιστα, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την έκθεση του κυρίου Βλάσαξ σε μεγάλη συντομία. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη εξ του είναι στο Στρασβούργο σήμερα, στο συνέδριο Νοτά ε, των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και μου ζήτησε να παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης εξ ονόματός του και να τονίσω ορισμένα βασικά σημεία. Πρώτον, είναι σαφές ε, σε όλους μας ότι η πολιτική συνοχή είναι σημαντική ε, οικονομική πηγή εισοδήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, μάλλον ε, τα θεσμικά όργανα, αλλά και τα κράτη-μέλη, οι πόλεις, οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση ε, θέλουν να προσελκύουν ε, επενδύσεις. Επίσης, για να τονώσουμε την οικονομία μας, θα πρέπει να αξιοποιούμε εκείνες τις εταιρείες που παρέχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Είναι περίεργο ότι ε, και οι μεγάλες εταιρείες παράγουν προστιθέμενη αξία και δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τους κοινοτικού πόρους. Οι επιχειρηματίες, οι εταιρείες μας δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και σύμφωνα με μια ε, ε, πρόσφατη έρευνα της Ernst Young, 33% των επιχειρήσεων ανησυχούν για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, 30% για τη φορολογία και 25% για την απασχόληση. Επίσης, η γνωμοδότηση τονίζει τη σημασία των πόλεων μας για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Ευκαιρίες επενδυτικές είναι πάρα πολλές, αλλά δεν προσελκύονται πάντα οι σωστοί επενδυτική εταιρία μας. Ε, χρειάζεται καινοτομία, χρειάζεται ε, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας για να τους προσελκύουμε. Προσπαθεί ο κύριος Βλάσακ να προτείνει τις καλύτερες λύσεις. Είναι πρόθυμος να ε, συναντηθεί στο Στρασβούργο με τους κοιόδης για να συζητήσει λεπτομέρειες και θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις για να τις διαβιβάσω στον κύριο Βλάσακ τα βασικά σας σχόλια και τις βασικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ο Ντέρεκ Βόν από τους Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και όλες οι γνωμοδοτήσεις και η παρούσα είναι πάρα πολύ σύντομη, γι' αυτό θα είμαι και εγώ σύντομο στα σχόλιά μου. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην προσέλκυση επενδύσεων. Είναι χαμηλή ανάπτυξη και ψηλή ανεργία και μάλιστα η απεργία η ενέργεια συγγνώμη, των νέων. Καλές οι προτάσεις νομοδότησης, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε ε, ε, επενδύσεις για την καινοτομία, για την κοινωνική ανάπτυξη, για τις υποδομές, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Γίνεται λόγος για τη σημασία των μεγάλων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επενδύσεις. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε και τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα των κοινωνικών εταιριών στην Ένωση. Όλοι έχουμε το ρόλο μας να παίξουμε και όλες οι εταιρείες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επίσης η γνωμοδότηση ε, μιλά για τη σημασία ε, της ε, πολιτικής συνοχής στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες πολιτική συνοχής και τα διορθωτικά ταμεία επιφέρουν ε, όφελος και για τις ε, ευημερούσεις περιοχές γιατί αναπτύσσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες και έτσι δημιουργούν αγορές ε, που θα απορροφήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πιο ανεπτυγμένων. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Επίσης γίνεται λόγος για κάποια από τα προβλήματα ως προς την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται λόγος για υψηλό δημόσιο χρέος και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα γιατί δεν έχουμε επενδύσεις, δεν έχουμε απασχόληση, δεν έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Είναι χαμηλή επένδυση στην υποδομή, στα προσόντα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναφερθούν στην έκθεση. Το τελευταίο σημείο ε, ε, συζητεί για, τη δυναμική των πόλεων. Το συζητήσαμε και προηγουμένως. Θα κάνουμε και τροπολογίες αλλά θα αξιοποιήσω και την ευκαιρία της συζήτηση με τον ο εισηγητή. Η κυρία Σισμένοβα δεν είναι εδώ. Ε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο ξανά, παρακαλώ. Εδώ είναι η κυρία Σισμένοβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. όχι. Η κυρία Μάνερ. Θα παρουσιάσω εγώ ε, τις απόψεις για το σχέδιο αυτό της γνωμοδότησης. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον συντάκτη η κυρία Χουσμένοβα ε, θεωρεί σωστά τα περισσότερα σημεία ε, συνάδουν με τη θέση της ομάδας μας. Η κυρία Σουσμένοβα θεωρεί και συμφωνεί με τον συγγήτη ότι η προσέλκυση των επενδύσεων είναι εκ των όνου κάνευ και μπορεί να υποστηριχθεί ε, και από την πολιτική συνοχή και τους στόχους Ευρώπης για το 2020. Προστιθέμενη αξία κάθε ευρώ που επενδύει ο δημόσιος τομέας προσελκύει περισσότερες επενδύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα στα έργα υποδομών και άλλα. Η προσέλκυση των επενδύσεων στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται σε κίνητρα που δίνονται επενδυτικά για να μπορούν οι περιφέρειες να δίνουν σωστά κίνητρα για να αυξηθούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Ε, στην τεχνολογία επίσης και στην τεχνογνωσία θα πρέπει να ενισχύεται αυτή με τη δημιουργία κέντρων, clusters, για να αυξάνεται η προσέλκυση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Η κυρία Χρυσμένοβα θέλει να τονίσει τη σημασία επίσης πολιτικής συνοχής για την έρευνα και την καινοτομία για την ευρωπαϊκή οικονομία και επίσης πιστεύει ότι οι επενδύσεις ε, στις υποδομές ε, τεχνολογίας, στην ευρυζωνικότητα και σε άλλες, καθώς επίσης και στο ανθρώπινο δυναμικό είναι κρίσιμες για να δημιουργηθεί ένα πιο, ε, ε, φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και προς τις επενδύσεις. Ευνοϊκό για τις επενδύσεις θα πρέπει ε, στόχος να είναι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί περίπου 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράγουν το 99% του τζίρου, ενώ απασχολούν πάνω από 2 τρίτα όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Καινοτομία λοιπόν, απασχόληση, κοινωνική συμπερίληψη, ε, φροντίζουν για όλα αυτά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν ε, μεγάλη πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας. Θεωρεί η ομάδα μας ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα βασικά από τη σκιώδη μας συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Σρέτερ. Um, Μάλιστα. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι η γενική μείωση των φορολογικών συντελεστών θα προσελκύσει επενδύσεις. Άλλα είναι τα σημεία. Αν υπάρχουν αρκετοί ειδικευμένοι εργαζόμενοι επιτόπου με τα σωστά προσόντα, εάν είναι σωστό το γενικότερο πλαίσιο και πεδίο. Δηλαδή, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ε, τους κατάλληλους εργαζομένους, είναι αρκετά ε, ελκυστική η περιοχή ε, σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τον πολιτισμό, γενικότερα δεν είναι μόνο το φορολογικό κίνητρο. Το βλέπουμε στις νέες χώρες ότι μπορεί να έχουν πάει οι εταιρείε εκεί ε, όσο έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά μετά από μια τριετία ή μια πενταετία αποχωρούν, γιατί έρχεται η επόμενη χώρα που μειώνει τους φόρους και είναι πιο ελκυστική. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Και δεν συμφωνώ με την έκθεση. Στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι ε, να τρέχουν οι εταιρείε από εδώ και από εκεί ε, και να κυνηγούν τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει να είναι σωστές ε, οι επιδοτήσεις για την επενδύση και τα κίνητρα, αλλά ε, να είναι σωστό και το πλαίσιο για να παραμένουν στο δυνικές και να επενδύουμε στους ειδικούς ε, εργαζομένους και πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό ηλιακό κλάστερ στην Ευρώπη, ανθεί η περιφέρεια μας, αλλά έχουμε τεράστια έλλειψη ειδικών εργαζομένων και γι' αυτό έχει σταματήσει η ανάπτυξη σχεδόν. Δεν μπορεί να συνεχίσει να ανθίζει γιατί δεν έχουν τους εργαζομένους που τους χρειάζονται να εργάζονται εκεί, να παράγουν και αυτό δείχνει ότι είναι αρνητική εξέλιξη και χρειάζεται νέα μεταρρύθμιση εκεί. Γι' αυτό με τους θεματικούς στόχους του 2020 είναι η σωστή προσέγγιση. Όχι απλώς λοιπόν φορολογικά κίνητρα. Αυτή θα ε, ήταν η σωστή κατεύθυνση. Και έτσι θα ήθελα την γνωμοδότηση. Θα την αλλάξω λίγο με τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Sean Kelly, please. Ευχαριστώ. Ο Σον Κέλλη. Κυρία Πρόεδρε, και πάλι η πολιτική συνοχής ε, είναι ένα βασικό θέμα και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αλλά ε, ε, υπάρχει και ένα άλλο βασικό επιχείρημα ότι ε, όσο αυξάνεται η ισχύς και η δύναμη των επιχειρήσεων τόσο πιο χρήσιμες είναι στην Ευρώπη γι' αυτό πρέπει να επενδύουμε στην Ευρώπη και αυτό που ελέγχθη είναι πολύ σωστό δηλαδή μέρος Τη στρατηγική στρατηγικής του 2020 αποβλέπει στην αύξηση τη χρηματοδότηση την οποία θα αφιερώσουμε στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη. Και αν αυτή η παραγωγή ε, δεν ε, ε, ολοκληρωθεί στην Ευρώπη, χάνουμε το χρόνο μας. Βλέπουμε ότι έχουμε τόσα νέα προϊόντα που παράγονται και ουσιαστικά παράγονται εκτός Ευρώπης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει να προσελκύσουμε την ελίτ, τους καλύτερους, όχι μόνο για να μείνουν στην Ευρώπη αλλά να τους διευκολύνουμε και με τις θεωρήσεις και τα λοιπά. Αν δείτε το ποσοστό των ε, βραβείων Νόμπελ στην Αμερική δεν είναι Αμερικανοί αλλά έχουν προσελκυστεί από τις συνθήκες. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο διότι όσο καλύτερη ποιότητα έχουμε σε ερευνητές τόσο περισσότερες ε, θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και τόσο τα περισσότερα ωφέλη θα έχουμε. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Τρεις παρατηρήσεις σύντομα. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις από πλευράς της δικής μας Επιτροπής έχουν δύο στόχους. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει βέβαια το αρχικό κείμενο της επί της ουσίας υπεύθυνης Επιτροπής. Πρώτος στόχος είναι να προσελκύσουμε επενδυτές και να δημιουργήσουμε σωστές συνθήκες για τους επενδυτές μέσω φορολογικών ρυθμίσεων, διευκολύνσεων κτλ. Και δεύτερον είναι τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ευρώπη. Για τον πρώτο τομέα δεν θέλω να κάνω τίποτα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι από άλλες επιτροπές. Για το δεύτερο κομμάτι Είναι σαφές ότι για τον κανονισμό με τον οποίο εργαζόμαστε έχουμε δύο θα έλεγα εξαιρέσεις. Καταρχάς έχουμε την εξαίρεση των παραγωγικών στοιχείων από μεγάλες επιχειρήσεις που θα απαγορεύονται αν θέλετε για το IDF και αν κατάλαβα καλά το κείμενο του Βλάσεκ αυτό θέλει. Πρέπει να απαγορεύσουμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις να επιδοτούνται για τα στοιχεία της παραγωγής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θέμα και δεύτερον για τις αναπτυγμένες περιοχές απαγορεύεται να χρηματοδοτούν τις βασικές υποδομές όπως τις μεταφορές, το περιβάλλον κτλ. Συνεπώς, προετοιμάζοντας ένα κείμενο, βλέπουμε ότι έχουμε μια αντίστροφη θέση σε ένα άλλο κείμενο. Εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια στοιχεία που έχουμε κάνει δεκτά στο παρελθόν. Ο Βανίστελ Ρόι έχει το λόγο. Συμφωνώ με τον Γιάννα Όρμπιχτ. Θα πρέπει να εισαγωγούμε κάποια καινοτόμα μέσα. Ε, μια μέθοδο ε, για το Περιφερειακό Ταμείο ιδιαίτερα, για πιο ευφυή ε, χρήση, για καλύτερη χρήση των εργαζομένων που να έχουν ε, περισσότερα προσόντα, να είναι πιο καλά εκπαιδευμένοι στην περιφέρεια. Να προσελκύσουμε τον κόσμο, αλλά όχι με τρόπο κατακαιρματισμένο, με ένα σωστό σύστημα. Για να έρχονται εταιρείε να εγκαθίστανται, ακριβώς επειδή ισχύουν ε, κάποιες προϋποθέσεις. Είναι μια ιδιαίτερη εδαφική διάσταση αυτή. Και να χρησιμοποιούμε διαφορετικά τους οικονομικούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας με δάνεια και με δραστηριότητες ε, όπου γίνεται ένας επιμερισμός του κινδύνου. Κατά τα άλλα καλή είναι η έκθεση, αλλά θα μπορούσαμε να τονίσουμε και το γεγονός ότι οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της τεχνολογίας προσφέρουν θαυμάσεις δυνατότητες σε περιφέρειες που απέχουν ίσως λίγο περισσότερο από τα κέντρα. Και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να είναι ελκυστικές, είναι start-up. Πολλοί νέοι θέλουν να αξιοποιήσουν όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν και μπορούν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται ότι το 40% των νέων θέσεων απασχόλησης θα έχουν σχέση με το διαδίκτυο. Να το δούμε αυτό πιο συγκεκριμένα και σε συνεργασία με τον Ούλγεχ. Έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα τελευταία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή μα και του συναδέλφου που ασχολήθηκαν με τη γνωμοδότηση τη ε, έκθεση που έχω αναλάβει να συντάξω για την ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Ποιος ήταν ο στόχος της έκθεσης ε, για τις ε, ανάγκες ανάπτυξης και βιώσιμης ανάπτυξης ιδιαίτερα της Ευρώπης έχουμε μιλήσει με πολλές αφορμές και, με πολλές, ε, και σε πολλές εκθέσεις τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και εδώ. Ο στόχος αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας είναι να τονίσει ότι η Ευρώπη παραμένει να, είναι ο πρώτος επενδυτικός προορισμός στον κόσμο αλλά απειλείται με τις ε, αναδυόμενες ε, αγορές οι οποίες έλκουν διεθνείς επενδύσεις και από αγορές που έχουν δυνατότητες να κάνουν ε, και από χώρες που έχουν δυνατότητες να κάνουν επενδύσεις στις ίδιες τις χώρες, άρα να μην εξάγουν αλλού τις επενδύσεις τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε, μας απασχολήσει πώς σε αυτή τη ε, ε, δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η Ευρώπη με τα δημοσιονομικά προβλήματα, με, τις, με τα θεσμικά της θέματα να αντιμετωπίσει και με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τον, διεθνή, τον ανταγωνισμό από άλλε χώρε πρέπει να, να, να, να αντιμετωπίσει τι αδυναμίε τη και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά τη για να μπορέσει να έλξει επενδύσει. ε, και να κρατήσει αυτή την πρωτοκαθεδρία που έχει του πρώτου προορισμού σήμερα, ο οποίο, επαναλαμβάνω, απειλείται από τι εσωτερικέ αδυναμίε τη και από τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Δεύτερο λόγο που με έκανε να πάρω την πρωτοβουλία αυτή τη έκθεση είναι ότι όταν λέμε ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτο προορισμό, μιλάμε σε ένα σύνολο. Και αυτό το σύνολο δημιουργείται από την ανταγωνιστικότητα κάποιων συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών. Δεν υπάρχει ισομέρεια στην κατανομή και στην έλξη επενδύσεων από όλες τις περιοχές. Άρα, πιστή στο στόχο της περιφερειακής συνοχής και σύγκλησης η Επιτροπή μας έχει κάθε λόγο να το αναδείξει αυτό το χαρακτηριστικό ότι πρέπει να δούμε πώς η έλξη των επενδύσεων κατανέμεται με ισομέρεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο τι κάνει ανταγωνιστική μια περιοχή. Δεν θα σταθώ στα θέματα που είπαν ήδη οι συνάδελφοι, ε, τα έχουμε τόσες φορές συζητήσει για το τι πρέπει να αξιοποιήσουν οι περιφέρειές μας, τους πόρους, θα έλεγα και τα συμπληρωματικά εργαλεία τη διευκολύνση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Συμπράξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα έχουμε πει με πολλές ευκαιρίες αυτά. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το, ότι οι, οι υποδομές, όχι μόνο οι, οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, αλλά και οι κοινωνικές υποδομές είναι πολύ σημαντικές για να κρατήσουν επενδύσεις και να έλξουν καινούριε. Και όταν λέμε επενδύσει εννοούμε και local και, από το, ε, και άμεσες διεθνείς επενδύσεις. Λοιπόν, οι υποδομές, κάθε είδους υποδομές, γιατί έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε μόνο λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια, αλλά είναι και οι κοινωνικές υποδομές, το φιλικό περιβάλλον υποδοχής των ξένων επενδυτών, ξένων εργαζομένων, η εκπαίδευση του, του ντόπιου προσωπικού, αλλά είναι δύσκολο όταν μια καινοτόμα επιχείρηση εγκατασταθεί κάπου να βρει αυτόματα ε, το όποιο προσωπικό δεν είναι αυτονόητο. Γι' αυτό η έκθεση τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης και της κινητικότητας προσωπικού. Άλλο σημαντικό θέμα είναι, το έθεσε ο κύριος Λούχαν, είναι το θέμα της έρευνας. Πώς η έρευνα διαχέεται και αξιοποιείται από όλες τις επιχειρήσεις σε όλες τις περιοχές. Εγώ συμπληρώνω ότι η παραγωγή της έρευνας είναι σημαντικό γιατί πάσχει σε αυτό το σημείο η ευρωπαϊκή έρευνα να εκπορεύεται από πάνω, από τα πανεπιστήμια, από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να παράγεται και local. Οι περιοχές έχουν σήμερα, όλες οι περιοχές έχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να παράγουν και ντόπια την έρευνά τους που πηγάζει από τις ανάγκες της αγοράς και συνεργάζεται με την αγορά. Είναι πολύ σημαντικό για να την αξιοποιήσει αυτόματα και η τοπική κοινωνία και, και η αγορά. Άλλο σημαντικό θέμα είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα δίνουν προστιθεμένη αξία σε αυτά που κάνει κάθε περιφέρεια. Φέρουν, ενώνουν τις ζωντανές, τις πλούσιες με τις φτωχές, τις απομονωμένες περιφέρειες. Δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα επενδυτικό μεγάλο στις, σε κάποιες περιφέρειες που δεν το έχουν από μόνες τους με το, στο πλαίσιο των εθνικών υποδομών. Ε, Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με την έκθεση την οποία συντάσσω και με την ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Όσο για την έκθεση του συναδέλφου κ. Βλάσπαρ είμαι πολύ ε, ευτυχής που έχει θίξει πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ θέλω να πω ότι ε, η έκφραση στην ε, παράγραφο 2 που λέει ότι δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα μοναδικό κριτήριο την ποιότητα και τη βιωσιμότητα ε, θεωρώ ότι η έκφραση δεν είναι επιτυχημένη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται μεγάλες επενδύσεις στι στις περιφέρειες αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα όλων των επενδύσεων, μικρών και μεγάλων. Δεν νομίζω ότι, ε, ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε από αυτά τα κριτήρια της μικρές, τι μεγάλες επενδύσεις. Ε, κάτι άλλο το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που η έκθεση δική μου ε, υποστηρίζει είναι ότι πρέπει ε, για τη συνοχή της Ευρώπης, για την συμπληρωματικότητα, για τον υγιή ανταγωνισμό να οδηγηθούμε σε μια σύγκληση και των οικονομικών και των φορολογικών και των κοινωνικών πολιτικών. δεν χρειάζεται να πω εδώ σε εσά ότι δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για μια ομοιόμορφη ε, οικονομική και κοινωνική πολιτική, αλλά αναφυσβήτητα η σύγκληση θα δώσει προστιθεμένη αξία στην Ευρώπη. Το άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πιο συντονισμένη πολιτική προβολής των πλεονεκτημάτων των περιφερειών μας. Ε, ταξιδεύω πολύ και εκτός Ευρώπης και έχω επαφή με μεγάλους επενδυτικούς φορείς, με ταμεία ε, επενδυτικά, με φαντς επενδυτικά, ακριβώς να δω πώς βλέπουν την Ευρώπη. Είναι μεγάλη σημασία για αυτούς η σταθερότητα της Ευρωζώνης και η στενή συνεργασία της Ευρωζώνης με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Θέλουν να δουν σε οποιαδήποτε περιφέρεια και αν έχουν στο νου τους να επενδύσουν, θέλουν να τη δουν σαν ένα μέρος ενός δυνατού συνόλου. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό η αξία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Γι' αυτό η εκπαίδευση και έρευνα είναι μεγάλη σημασία για τις περιφέρειες, διότι αισθάνονται οι ξένοι επενδυτές ότι παντού στην Ευρώπη υπάρχει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό, το ποιοτικό και το ανταγωνιστικό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε την Ευρώπη. Η ενιαία αγορά είναι ένα μεγάλο, ε, μεγάλο δημιούργημα το οποίο δίνει προστιθεμένη αξία σε κάθε προσπάθεια περιφέρειας. Αυτή η ενιαία αγορά νομίζω ότι πρέπει να προβληθεί. Δεν, είναι, δεν πρέπει οι επενδυτέ να σκέφτονται μόνο τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, ε, την Ελλάδα όταν, κάνουν ε, όταν σκέφτονται να κάνουν επενδύσεις. Πρέπει να σκέφτονται τη Γαλλία, την Πολωνία κτλ. Αλλά στο πλαίσιο της ενιαία αγοράς. Έχουμε όπλα τα οποία α, δίνουν, ο σύνολο, έχουμε κατακτήσει όπλα τα οποία δίνουν προστιθεμένη αξία στην κάθε περιφέρεια. Και αυτά πρέπει και να τα ενισχύσουμε, ενισχύοντας τη μεγάλη, την ενιαία αγορά, τη σταθερότητα, την δημοσιονομική, και να τα προβάλλουμε και μέσα στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που φέρνει η έκθεση σε σχέση με αυτά που έχουν πολλές φορές τονιστεί και από τη δική μας Επιτροπή και από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Είναι σημαντικές για την γνωμοδότηση. Νομίζω ότι ο κύριος Βλάσεκ θα μπορέσει να τις λάβει υπόψη του όλες και να καταλήξουν σε μια σωστή λύση. Τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 29 Μαρτίου 12 μεσημβρινή. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν το συζητήσαμε. Είναι Νούνο Τεσέιρα. Δεν έχουμε όμως χρόνο, οπότε κανονικά θα πρέπει αύριο κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Θα δούμε όμως Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν το λόγο και οι σκιώδεις εισηγητές και τα λοιπά δεν θα είναι... Ε, εκτός αν δεν υπάρχει βέβαια κάποιος που θέλει το λόγο, οπότε μπορούμε να βάλουμε μόνο την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Αν δεν υπάρχουν ομιλητές οι οποίοι θέλουν να πάρουν το λόγο, μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας και απλά να βάλουμε την προθεσμία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία ήρθα. Αυτό ίσως σας μπέρδεψε λίγο στην τήρηση της σημερίσίας διάταξης. Θα ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει ανάγκη από μια γρήγορη και απαραίτητη μεταρρύθμιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία της αηφορίας, τα στοιχεία της οικολογίας, τα πολιτιστικά στοιχεία και είναι απαραίτητο επίσης να υπάρξει και ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 όπως επίσης και καλύτερο συντονισμό των πολιτικών που πλαισιώνουν τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει περισσότερες ευθύνες στα πλαίσια της διαχείρισης της αλίας και μέσω της επικουρικότητας θα πρέπει να υπάρξει όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή ε, και των περιφερειακών αρχών και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Αυτό είναι βασικό για να υπάρξει μια μεταρρυθμισμένη πολιτική που θα βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της στρατηγικής επαναλαμβάνω 2020. Υπολογίζω στην στήριξή σας και ελπίζω ότι με τη συνεργασία όλων σας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών και πάλι 29 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Και έτσι εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση επιτροπής, ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ αποχωρήσετε όσο μπορείτε πιο σύντομα για να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. We working in these letters to the Σε μισή ώρα εδώ στην αίθουσα θα συνεδριάσει η ομάδα εργασίας με τη Δανική Προεδρία θα μας ενημερώσει η Προεδρία για την κατάσταση των πραγμάτων και την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Παρακαλώ όσοι φεύγετε να ξανάρθετε στις 6.30.